Καλημέρα σας. Θα αρχίσουμε τις εργασίες μας. Άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και περνάμε στο πρώτο θέμα απευθείας. Εκθεσή του κυρίου Στόλοζαν για την αμοιβαία συνδρομή για την ίσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα. Σας δίνω το λόγο, κύριε Στόλοζαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το σχέδιο οδηγίας είναι εξαιρετικά τεχνικό. Τίθενται διάφορα σημαντικά ζητήματα. Αυτή η νέα οδηγία χρειάζεται λόγω της κινητικότητας του κεφαλαίου και του εργατικού δυναμικού. Χρειάζεται λοιπόν αμοιβαία συνδρομή ανάμεσα στα κράτη-μέλη για την εισπράξη απαιτήσεων σχετικά με κάποιους φόρους. Το φαινόμενο αυτό έχει αυξανόμενη σημασία. Το 2003 είχαμε 3.000 αιτήσει και περάσαμε σε άνω των 8.000 το 2008. Δυστυχώς η αποτελεσματικότητα για την ίσπραξη απαιτήσεων είναι εξαιρετικά χαμηλή. Κυμαίνεται στο 5% περίπου των ε, απαιτούμενων ποσών. Βλέπετε την πρόταση της νέας οδηγίας. Και συνοψίζοντας ε, θα έλεγα ότι πρόκειται για τη διεύρυνση καταρχάς ε, του πεδίου εφαρμογής σχετικά με την αμοιβαία σύνδρομη για να καλύψει και τις υποχρεωτικές εθνικές ε, ασφαλιστικές εισφορές, αποκλείοντας όμως τα πρόστιμα και τις χρηματικές ποινές σε ποινικέ διαδικασίες. Η οδηγία καλύπτει επίσης την εισαγωγή ομοιόμορφων εργαλείων που επιτρέπουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων Επίσης ένα συγκεκριμένο έντυπο για την κοινοποίηση των εγγράφων και υπάρχει και μια άλλη πρόταση χάρη στην οποία εκπρόσωποι των κρατών μελών μπορούν να συμμετάσχουν ένεργα σε διοικητικές έρευνες που διεξάγονται στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους. Το τελευταίο σημαντικό σημείο είναι ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών ή εγγράφων πρέπει να κοινοποιείται με ψηφιακό τρόπο χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό δίκτυο. Όπως σας είπα, το σχέδιο οδηγίας φαίνεται πάρα πολύ τεχνικό. Διάφορα ζητήματα δε ακόμη συζητώνται σε διάφορα κράτη-μέλη, σε συνεδριάσεις που είχα με διάφορους υπαλλήλους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπους των κρατών μελών έμαθα πως συνεχίζονται οι συζητήσεις ούτως ώστε να συμπεριληφθούν και υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές στο πεδίο εφαρμογής της αμοιβαίας συνδρομής. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριληφθούν αυτές οι εισφορές, δηλαδή τάσομαι υπέρ της θέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συζητείται επίσης η αποδοχή της παρουσίας των εκπροσώπων κάποιου κράτους μέλους στις ε, διοικητικές υπηρεσίες ενός άλλου κράτους μέλους και τη συμμετοχή τους σε διοικητικές έρευνες άλλου κράτους μέλους. Ε, κάποια κράτη-μέλη ανθίστανται σε αυτή την πρόταση, αλλά πάλι υποστηρίζουν αυτή την πρόταση. Εγώ υποστηρίζω τη συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, διότι θεωρώ ότι λόγω της ολοκλήρωσης ε, των κρατών μελών και της ε, ενιαίας αγοράς και της αυξανόμενης κινητικότητας του κεφαλαίου και του εργατικού δυναμικού καθιστούν απαραίτητη την ολοκλήρωση και σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει επίσης ε, πρόταση μέσα στο σχέδιο οδηγίας για ένα αρχικό εργαλείο στο ετών κράτος μέλος συνήθως χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους έγγραφα στον τομέα της δικαιοσύνης. Η αίτηση που προβλέπεται στην οδηγία προβλέπει αυτά τα έγγραφα, αυτά τα εργαλεία να περιοριστούν σε ένα ομοιόμορφο έντυπο που θα αποστέλλεται στο άλλο κράτος μέλος, προσού η αίτηση, έχω λάβει διάφορα σχόλια που ζητούν να μην είναι απαραίτητη αυτή η χρήση του ενιαίου εργαλείου, του ενιαίου εντύπου, για τον εξής λόγο. Ενίοτε σε κάποια κράτη-μέλη τα αρχικά έγγραφα που εκδίδονται ε, στον τομέα της δικαιοσύνης πρέπει να παραμένουν στην επικράτεια του κράτους μέλους και οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες ε, επιθυμούν τη διατήρηση αυτών των αρχικών εγγράφων και τελειώς πρέπει να τρέχουν στους συμβολεογράφους για να επικυρώσουν τα αντίτυπα κτλ. Και στην εκδίκαση μην ξεχνάτε ότι πρέπει να υποβάλλονται τα πρωτότυπα έγγραφα. Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Με τα χαράς να ακούσω τις προτάσεις και τα σχόλια των μελών, ώστε να οριστικοποιήσω το σχέδιο της έκθεσης και να ε, το υποβάλουμε ταχύτερο δυνατόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στόλζαν. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους κοιόδης από τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Βάινγουοκ ε, από τους Σοσιαλιστές ε, θα πάρει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έγγραφο εργασίας που μας διαβίβασε. Προκύπτουν σαφώς τα ζητήματα που τίθενται μέσα σε αυτό το σχέδιο οδηγίας. Συμφωνώ μαζί του σχετικά με την πρόοδο που συνιστά η συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογή του σχεδίου οδηγίας των υποχρεωστικών ασφαλιστικών εισφορών και την δυνατότητα των υπαλλήλων του σε κράτου μέλους να συμμετάσχουν στη διεξαγωγή έρευνα σε άλλο κράτο μέλο. σχετικά με την υποβολή του πρωτότυπου εγγράφου μαζί με το ε, ομοιόμορφο έντυπο, νομίζω ότι υπάρχει παρανόηση. Δεν πρόκειται περί αυτού. Ένα επικυρωμένο αντίτυπο, γνήσιο αντίτυπο του πρωτότυπου εγγράφου, περί αυτού πρόκειται. Οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω θα μπορέσουν να μα καθησυχάσουν στη συνέχεια σχετικά με αυτό το θέμα. Δύο σημεία μου φαίνεται ότι έχουν μεγάλη σημασία για να δώσουμε εγγυήσει για την αποτελεσματικότητα τη οδηγία. Καταρχάς ένα τεχνικό θέμα. Φαίνεται ότι η πρόταση ε, έχει κάποιες ελλείψεις σε επίπεδο εγγυήσεων για τις προθεσμίες, ιδιαίτερα για την περίοδο παραγραφής των διαδικασιών. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί πολλές από τις διαδικασίες δεν ολοκληρώνονται μόνο και μόνο λόγω των καθυστερήσεων. Το επόμενο θέμα είναι λιγότερο συνενετικό θα έλεγα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει δύο πολύ περιοριστικά μέτρα. Το πρώτο θεωρεί ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη δεν μπορεί να γίνει παρά για τις περιπτώσεις απάτης άνω των 10.000 ευρώ. Τη στιγμή που το Κοινοβούλιο εκφράζεται υπέρ της ανταλλαγής της αυτόματης φορολογικών πληροφοριών, εκτός από την κυρία Λούλινγκ βέβαια, θα ήταν λυπηρό να μείνουμε σε ένα τόσο υψηλό όριο και δίδει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αρνηθούν την συνεργασία τους και την ανταλλαγή πληροφοριών εφόσον θεωρούν ότι αυτή θα θέσει σε κίνδυνο ένα βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό μυστικό ή θα ήταν τέτοια φύσεως που θα έφυγε την δημόσια τάξη και την ασφάλεια του συγκεκριμένου κράτους. Αυτές οι προβλέψεις ε, ε, υποθέτουν ότι υπάρχουν ορισμένοι απατεώνες θα έλεγα, ίσως κάποιες τράπεζες, ίσως κάποια άλλα πιστοτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν ασυλία. Αυτό είναι νομίζω ε, κατά του κώδικα κοινή συμπεριφοράς. Η κρίση χτυπάει πολύ περισσότερο τους πιο εύθραστους από τους συμπολίτε μας και γι' αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε αυτή την αρχή της ισότητας μπροστά στη δικαιοσύνη. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι η έκθεση του κυρίου Στόλογιαν είναι μια εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Χουανγνόκ. Και τώρα το λόγο έχει κύριο κύριος Ολέσμιτ από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Νομίζω ότι αυτό το έγγραφο εργασίας είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ δύσκολα τα θέματα. Το θέμα είναι τεχνικό, ε, είναι και θέμα αρχών όμως και ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Ευρώπη περί τα φορολογικά αν ξεστομίσει εδώ κανείς τη λέξη φορολογία, θα αρχίσουν να οριάζουν διάφοροι συνάδελφοι στην Επιτροπή μας. Αυτές τις μέρες έχει αλλάξει λίγο το πνεύμα και το κλίμα και ίσως γι' αυτό ε, ε, έχει πιο ευνοϊκό και θετικό ύφος στο εγγραφό του εισηγητής. Διότι γνωρίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ όλων των κρατών μελών για να αρχίσει η διαδικασία αυτή καν. Και θα ήθελα να πω από πλευρά μα, ενώ τη πολιτική μου ομάδα, ότι εμεί συμφωνούμε με όλα αυτά που λέτε και θα σα υποστηρίζαμε. Αλλά δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Ε, όπως είπε ο συνάδελφος, πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα διάστημα που είναι ευκαιρία. Ξέρουμε όμως τις διαφορετικές απόψεις και πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα στο παρελθόν τουλάχιστον. Διαβάζοντας και το έγγραφο σας και την οδηγία, θα έλεγα ότι εσείς τονίσατε την και τα προβληματικά σημεία της οδηγίας το θέμα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, ε, αμοιβαία συνδρομή, συμφωνώ. Αλλά κάποια επιχειρήματα θα πρέπει να βρούμε εις βάρος. Και η παρουσία υπαλλήλων κράτους μέλους στις εφορίες ή στις υπηρεσίες άλλων κρατών Και αυτό είναι επίμαχο. και η εφαρμογή και ε, στα υποψήφια κρατημέλη. Εδώ διστάζετε λίγο στα σχόλιά σας. Και μπορεί να έχετε και δίκιο. Παρόλο που υπάρχουν μερικά προβλήματα, οι προτάσεις είναι πολύ καλές και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πρόθυμη να ανταλλάσσει και πληροφορίες και να κάνει κάτι. Ξέρουμε το πρόβλημα με την οδηγία για τις καταθέσεις και όλες τις συζητήσεις αυτές που έγιναν, αλλά τελικά η θέση σήμερα αλλάζει. Γενικά συμφωνούμε και εσείς και εγώ ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ καλή. Μπορεί βεβαίως να τροποποιηθεί σε κάποια άρθρα της, αλλά γενικά νομίζω πρέπει να υποστηριχθούν. Γενικά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει συνένεση σε αυτά τα θέματα και μεγάλη πλειοψηφία να περνούν. Αλλιώ είναι μάλλον σχεδόν αδύνατο. Καλή τύχη λοιπόν κύριε Σιγητά μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σμιθ ο εκπρόσωπος ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ο κύριος Βαντεμπέρκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το θέμα για τη βελτίωση ε, της συνδρομής σε θέματα φορολογικά και άλλα είναι τμήμα της πρότασης για τη βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν θέλουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την απάτη, θα πρέπει να ε, ε, έχουμε απέτηση και ίσπραξη των φόρων εκεί που δεν συλλέγονται. Και το δικαστήριο λέει ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να ε, θέτουν προσκόμματα δικαιολόγητα στη διάφορη, στη, στην ελεύθερη κυκλοφορία. Έστω και αν πρόκειται για φόρους αλλά τα κράτη θα πρέπει να προχωρούν λέει, σε ε, πιο αποτελεσματική συνεργασία για την ίσπραξη ε, των απαιτήσεων που έχουν σχέση με φόρους. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες ε, της πρότασης, διότι ο συγητής το έκανε πάρα πολύ καλά και με πολλές λεπτομέρειες. Θα ήθελα μόνο να απαντήσω με μια διευκρίνηση στην ερώτηση που έγινε για τον ενιαίο τίτλο. Σύμφωνα με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός από τον τίτλο αυτό θα πρέπει να, να στέλνετε και ο αρχικός τίτλος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Τι θα πρέπει να στέλνουμε ως πληροφορίες. Και τα δύο. Είναι ηλεκτρονική η μορφή αποστολής των πληροφοριών, δεν είναι έγγραφο, όπως και η αίτηση και ε, η ομοιόμορφη ε, μορφή του εγγράφου, αλλά μπορεί να είναι και ακριβές αντίγραφο ε, του κειμένου που υπάρχει στη χώρα η οποία ε, απευθύνει το αίτημα. Ακριβές πάντα αντίγραφο όμως και με βεβαιωμένη την υπογραφή στην εκτελεστική δεν νομοθεσία, σε εφαρμοστικές διατάξεις, ισχύει ε, και σήμερα. Όταν στέλνουμε έγγραφα, και αυτά είναι αντίγραφα, μπορούν να θεωρηθούν ακριβή αντίγραφα και να θεωρηθούν γνήσια και να ισχύουν σαν να ήταν τα πραγματικά έγγραφα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγε να στέλνουμε και το πρωτότυπο για να υπάρχει ακριβής ενημέρωση για το μήνυση πραχθέντα φόρα. Και κανονικά ο φορολογούμενος θα πρέπει εκ των προτέρων να έχει λάβει το γνήσιο αρχικό κείμενο γιατί η αίτηση για αμοιβαία συνδρομή έρχεται σε απότερο στάδιο όταν δεν θα ε, έχει καταβάλει το φόρμα του αναλογή. Δηλαδή θα έχει πάρει πρώτα το καθαριστικό ο ενδιαφερόμενος και μετά ακολουθεί όλη αυτή η διαδικασία. Εφόσον όμως υπάρχει ακριβές αντίγραφο βεβαιωμένο, είναι σαν να έχουμε το ε, πρωτότυπο. Ευχαριστώ. Θέλετε να ε, κάνετε τις τελικές σας παρατηρήσεις. Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έκαναν προτάσεις, συστάσεις χρήσιμες. Νομίζω ότι οι παρατηρήσεις σας ε, σαφώς και μπορούν να πάρουν τη μορφή τροπολογιών θα σας παρουσιάσω πλέον το σχέδιο εκθέσεως μόλις το ετοιμάσω και εκ νέου απλά θα σας ευχαριστήσω σε αυτή τη φάση για την προσπάθειά σας. Νομίζω ότι η οδηγία αυτή είναι κάτι που χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Στολογιάν. Ολοκληρώνεται η συζήτηση για το σημείο αυτό της μέσης διάταξης και ανοίγουμε το επόμενο που είναι η έκθεση της πολιτικής ανταγωνισμού 2008. Η συγκήτρια είναι η κυρία Σόφι Νετβέλτ. Έχετε το λόγο. Um, yes, thank you. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη στην πρώτη παρουσίαση που θα κάνω για την έκθεση για την πολιτική του ανταγωνισμού. Στην προηγούμενη την είχε κάνει ο Τζόναθαν Evans. Να πω κάτι για τη διαδικασία και κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Ιδιαίτερα για την λεγόμενη διοργανική συνεργασία. Η έκθεση καλύπτει μία μεγάλη σειρά θεμάτων που θα χαρακτήριζα διαφορετικά μεταξύ τους και εγώ προσπαθώ να καταλήξω σε ένα κείμενο το οποίο να συνιστά ένα σαφές συνεκτικό πολιτικό μήνυμα και να μην είναι ένας απλός κατάλογος επιθυμιών ή αγορών. Ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει ένα τέτοιο μήνυμα ισχυρό. Αυτό μάλιστα πρέπει να γίνει γιατί μιλάμε για μια σύσταση αν θέλετε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι δεν θα πρέπει αυτή η ετήσια δήλωση ε, να είναι στην ουσία μια απλή ιεροτελεστία. Βλέπω ότι ο κύριος Φέμπερ έχει ενθουσιαστεί με αυτά που λέω αλλά να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτά τα οποία λέμε γιατί αλλιώς θα χάνουμε το χρόνο μας. Επανέρχομαι σε κάποιες από τις συστάσεις που έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια και οι οποίες δεν έχουν τύχει κατάλληλη συνέχεια και εφαρμογής. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει λίγο εδώ να κάνει κάτι. Υπήρξαν κάποιες ε, μελέτες τομεακές οι οποίες ζητήθηκαν, τις οποίες δεν προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μπορεί να έχει σωστούς λόγους που δεν έκανε κάτι τέτοιο, αλλά από την άλλη παραμένουν σε εκκρεμότητα. Θα ήθελα επίσης να βραχύνω χρονικά τη διαδικασία και να ζητήσουμε την αποδοχή της συγκεκριμένης έκθεσης από την Ολομέλεια τον μήνα Μάρτιο ελπίζοντας ότι έτσι θα επηρεάσουμε κάποιες από τις αποφάσεις που εκκρεμούν. Τυχαία λίγο θα σας δώσω κάποια από τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η έκθεση. Είναι σαφές ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται και οι τίτλοι που περιλαμβάνονται είναι πάρα πολλοί καλύπτονται τομείς όπως οι κρατικές επιδοτήσεις, οι κρατικές βοήθειες. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς κρατική βοήθεια έχει δοθεί στα πλαίσια των προγραμμάτων ανάκαμψης των οικονομιών των χωρών της Ένωσης. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε επίσης ποια είναι τα αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις αυτές να δούμε αν υπήρξαν κάποια προβλήματα, κάποιες συνέπειες, κάποια στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, ίσως ναι, ίσως όχι τι ποσοστό της κρατικής βοήθειας δόθηκε για την λεγόμενη πράσινη ανάκαμψη. Αυτή ήταν μία από τις προϋποθέσεις η οποία θα χαρακτήριζε την μορφή αυτή βοήθειας προς τον τομέα της βιομηχανίας να σχολιάσουμε λίγο τις στρατηγικές εξόδου από την κρίση και να μην τα δούμε αυτά μόνο στον προηγούμενο χρόνο, στην χρονιά δηλαδή που διανύουμε, αλλά να δούμε και το τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον, να δούμε τι πλαίσιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της χορήγησης βοήθειας προς τομείς άλλους του τραπεζικού. Αυτά είναι ο πυρήνας της ε, έκθεσης. Άλλοι τομείς είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις antitrust όπως επίσης και οι ρυθμίσεις των τομέα συνενώσεων συγχωνεύσεων εταιριών. Αυτά έχουν καλυφθεί και από προηγούμενες εκθέσεις, όπως η Λευκή Βίβλος που είχε προηγηθεί Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία συνδέονται με τις νομοθετικές ρυθμίσεις ε, ε, μαζικών ή συνολικών απαλλαγών και εξαιρέσεων σε τομείς όπως ο ασφαλιστικός. Υπάρχει επίσης η αναθεώρηση του κανονισμού 1-2003 Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη εδώ θα ήθελα να θέσω κυρίως το θέμα των προστήμων τα οποία επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και να συζητήσουμε για να δούμε αν πιστεύουμε ότι η βάση για τον υπολογισμό των προστήμων είναι η σωστότερη. Αυτή που χρησιμοποιείται δηλαδή είναι σωστή. Και ίσως ένα τελευταίο σημείο είναι η αναθεώρηση του κανονισμού για τις συγχωνεύσεις και υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία προκαλούν προβλήματα όπως το εάν επιθυμούμε να αναθεωρήσουμε κάποιους από τους κανόνες που ισχύουν σχετικά με το ποια αρχή θα ασχολείται με ορισμένες περιπτώσεις αν θα, το σύστημα το οποίο κατανέμει τις αρμοδιότητες από τη μία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την άλλη στις αρμόδιες εθνικές αρχές για τον ανταγωνισμό είναι ικανοποιητικό. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερο θέματα από πλευρά των συναδέλφων, να ανταλάβω υπόψη μου. Θα προετοιμάσω το προσχέδιο ίσως και την επόμενη εβδομάδα να είναι έτοιμο για να το στείλω στη μετάφραση. Και τώρα θα πρέπει η Γραμματεία να επιβεβαιώσει αυτό που θα πω, ίσως να γίνει δυνατόν η συζήτηση να λάβει ε, χώρα την 1η ή τη Δευτέρα Δεκεμβρίου να, να δεχθούμε τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο την συγκεκριμένη έκθεση σε επίπεδο επιτροπής έτσι ώστε να καταλήξουμε τον μήνα Μάρτιο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Thank you very much, ε, Ευχαριστώ πολύ Σοφή. Τώρα, πρώτος που έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Μπούλμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο σκιώδης ηγητής μας, ο Αντολίν Σάντσες Πρεσέντο, ε, είχε σοβαρή ανηλυμένη υποχρέωση και κολλείεται σήμερα παραστή. Πάντως υποστηρίζει τη γραμμή της ε, εισηγητρίας και προτίθεται να συνεργαστεί μαζί της. Χαίρεται για την ανταλλαγή απόψεων. Και κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον σκιώδη μας εισηγητή και για την ομάδα μας, γιατί αυτή τη γραμμή θα ακολουθήσουμε στη σημαντική τότε έκθεση, είναι να πούμε ότι αυτό τον καιρό που έχουμε τη χρηματοοικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση χρειάστηκε και ε, χρειάζεται ακόμα μαζική κρατική παρέμβαση. Αλλιώς δεν μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία και θα πρέπει να προσέξουμε ακριβώς αυτό το λόγο να μην έχουμε στρεβλώσει ανταγωνισμού. Αυτό είναι το σημαντικότερο λοιπόν και για τον συνάδελφό μου και για την ομάδα μας και γύρω από αυτό θα διαρθρωθεί ολόκληρη η ε, πρότασή του σε συνεργασία με την κυρία Νιτβέλτ. Ε, βέβαια για ε, την καταπολέμηση των καρτέλ τα στοιχεία Ε, λέγουν ότι οι ζημίε ανέρχονται ε, σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ και πλέον. Το ξέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό και θα πρέπει να κινητοποιηθούμε για να το αντιμετωπίσουμε. Καλό είναι λοιπόν να συζητάει το Κοινοβούλιο και να συνεννοείται για την πολιτική ανταγωνισμού. Η πολιτική καταπολέμηση των ε, συνεννοήσεων και κατά τον τραστ και τον καρτέλ είναι σημαντική γιατί έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αποζημίωσή τους. Υπάρχει και θέμα της εσωτερικής αγοράς για την ενέργεια και ο συγητής μας, ο συγητής, χαίρεται που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται και με ε, τον κλάδο των τροφίμων και ιδιαίτερα των γαλακτοκομικών ε, για να μην υπάρχει δεσπόζουσα θέση κάποιων ολιγοπολίων στην αγορά και ε, συνεννοήσεις για τις τιμές εις βάρος του τελικού καταναλωτή. Αυτά θα σας τα πει και ο ίδιος ε, σε επόμενη ευκαιρία όταν θα είναι παρόν. Ευχαριστώ κύριε Μπούλμα. Και τώρα το λόγο έχει ο σκιώδης ηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κ. Σφάπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω και ο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελα βεβαίω να ευχαριστήσω και την κυρία Ενετφέλτ και τον κύριο Μπούλμαν που εκπροσωπεί τον κύριο Σάντσε Πρεσέδο. Συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό και υποστηρίζω και εγώ τις ε, προτάσει. Τώρα, ε, στο δίκαιο ανταγωνισμού και στην καταπολέμηση των καρτέλ είμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση μεταβατική. Το είπε και η κυρία Ενετφέλτ, έχουμε νέο κοινοβούλιο και προσεχώ νέο επίτροπο. Το 2003 στον αντίστοιχο κανονισμό για την καταπολέμηση των καρτέλ είχε πει ότι σε έξι χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έξι χρόνια θα ε, τον αναθεωρούσε. Και χαίρομαι. για την έκθεση αυτή, αλλά τώρα δεν έχουμε αρκετό χώρο μετά που αποφάσισαν συντονιστεί και η Γραμματεία για εκθέσει ιδία πρωτοβουλία. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ελέγχονται τα καρτέλ ε, για την προστασία των καταναλωτών και το έχει συμπεριλάβει και στην πρότασή της. Η ετήσια έκθεση λοιπόν του 2008 είναι η σύνοψη της μεταβατικής αυτής κατάστασης που ζούμε. Το χρονοδιάγραμμα που μας προτείνει η κυρία Ινετβέλτ νομίζω ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξο. Αν θέλουμε να έχουμε στόχο την παρακολούθηση και τη συνέχεια και κάποιων άλλων εκθέσεων που έχει εγκρίνει η Επιτροπή μας, όπως η έκθεση του Τζόναθαν Εύαν στο παρελθόν από το Λαϊκό Κόμμα. Πάντως, εκφράζω την προθυμία της ομάδας μας να συνεργαστούμε και η έκθεση του 2008 Μόνο ακροθυγό αναφέρεται στις δυσκολίες της οικονομίας και στην κρίση που είπε και ο κύριος Μπούλμαν, γιατί αυτές φάνηκαν σε όλη του τη διάσταση, στη μεγαλύτερη διάστασή του στα τέλη του 2008. Εγώ ε, θα ήθελα να αναφερθώ στον κανονισμό 1 του 2003 γιατί για τα πολέμηση των ε, καρτέλ ε, και έρχομαι στο πρώτο ερώτημα. Το είπε και η συγκεκριά τι γίνεται με το σύστημα της συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς διαρθρώνεται αυτή η συνεργασία. Μέχρι τώρα ήταν το λεγόμενο one-stop shop όπου κανείς απευθύνεται σε μία υπηρεσία. Υπάρχει δυσκολία όμως λειτουργίας Αυτό που μα ενδιαφέρει στην Ευρώπη είναι το ελεύθερο εμπόριο, το δίκαιο εμπόριο, αλλά και ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και θέλουν να είναι νομοταγεί και να τηρούν τους κανόνες. Στη συνέχεια, τι γίνεται ε, στη συμμόρφωση, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να δίνουμε την ευκαιρία στις ε, επιχειρήσεις που θέλουν και τηρούν τις ευρωπαϊκές διατάξεις να ορθοποδήσουν. Υπάρχουν μεμονωμένες εταιρείε που κυριαρχούν στην αγορά και έχουν δεσπόζουσα θέση σε κάποια κράτη-μέλη. Εδώ νομίζω θα πρέπει τα κράτη να έχουν τη ε, δυνατότητα να δρουν στα πλαίσια της επικουρικότητας και αν θέλουν να επιβάλλουν πιο αυστηρές κυρώσεις από ό,τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνουν. Τι γίνεται επίσης με το σημείο 11 για την αποκάλυψη ε, καρτέλ και τις βασικές μαρτυρίες και τι γίνεται με το θέμα των ε, συλλογικών αγωγών. Μήπως ο καλύτερος δρόμος ε, ε, είναι να προχωρήσουμε προς το δρόμο της καταγγελίας για την αποκάλυψη των καρτέλ και όχι στις συλλογικές αγωγές. Δηλαδή κάποιος που θέλει να αποκαλύψει μια τέτοια στρεβλή πρακτική και ένα καρτέλ μπορεί να διστάσει γιατί στη συνέχεια ορισμένοι καταναλωτές θα ε, οργανωθούν και θα προσφύγουν συλλογικά στη δικαιοσύνη και αυτό θα είναι και εις βάρος. Τώρα τι γίνεται με τα πρόστιμα είναι πολύ υψηλά τα ποσά, έχουν αποτρεπτική ισχύ και μεγάλη που τη χρειαζόμαστε, δεν χωράει καμία αμφιβολία, αλλά υπάρχει οικονομική αναλογικότητα. Μήπως είναι δυσανάλογα, μήπως έχει εκφυλιστεί το σύστημα και η βασική ιδέα της διαδικασίας είναι να ελέγχει κιόλας το δικαστήριο ότι θα καταβάλλονται τα πρόστιμα. Εγώ δεν θέλω να μειωθούν τα πρόστιμα για τα καρτέλ, αλλά να έχουμε και στο μυαλό μας μια τάξη μεγέθους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες όταν ανήκουν σε ένα καρτέλ, σε ένα ολιγοπόλιο, εξαρτώνται 100% για τον τζίρο τους ε, ε, από αυτή τη σύμπραξη. Και όταν ε, τους επιβάλλεται τέτοιο μεγάλο πρόστιμο, γονατίζουν. Οι μεγάλες εταιρείες, ε, τα μεγάλα καρτέλ δεν έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα πρόστιμα γιατί είναι κολοσσοί και μπορούν να επομιστούν αυτό το κόστος. Θα πρότεινα να το συζητήσουμε με την εισηγήτρια μήπως χρειαστεί να οργανώσουμε και καμία ακρόαση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σουάμπ. Ο κύριος Λάμπερς. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί σοφοί. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, για αυτή την έκθεση. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι σοφή που θες να είσαι προσγειωμένη στο έδαφος και να υπάρχει και συνοχή σε σχέση με το παρελθόν. Όχι άλλη μια έκθεση μετά από μια σειρά εκθέσεων που ουσιαστικά δεν πολύ χρησιμοποιούνται. Το εκτιμούμε αυτό. Τώρα, κάποιες παρατηρήσεις. Δεν θέλεις shopping list, μας είπες. Ε, θέλεις ε, να υπάρχει μια έκθεση σχετικά με τη συνοχή αν όμω θέλουμε να έχει βάρος η έκθεση πρέπει να αντανακλά την πραγματικότητα που επικρατεί σε διάφορους κλάδους. Τι εννοώ. Αυτοκινητοβιομηχανία. Πρέπει να προσέξουμε γιατί τα συστήματα κρατικών ενισχύσεων που έχουν θεσπιστεί και εδώ συμφωνώ μαζί σου ενδεχομένως οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Το πιο σημαντικό όμως είναι το εξής μήπως έχουμε περιέλθει σε μια θέση τώρα όπου ε, κάποιοι ελάχιστοι φορείς ε, ελέγχουν τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές ε, ποιοι είναι οι προμηθευτές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως επιτοπλίστων και ε, τους ασκείται μεγάλη πίεση από αυτούς τους μεγάλους παίκτες της αγοράς και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς ε, έχει η κατάσταση στην αγορά. Δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα υγιής η διαπραγματευτική ε, δυνατότητα που έχουν οι προμηθευτές σε σχέση με τους μεγάλους παίκτες δεν είναι πάρα πολύ καλή και αυτό χειροτερεύει τα τελευταία χρόνια. Ε, για τη λιανική πώληση, τους τελευταίους μήνες ε, παρατηρούμε ότι υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός ανάμεσα στους ε, λιανοπολιτές αλλά και πάλι τίθε το ζήτημα της ισχύω που έχουν σε σχέση με τους προμηθευτές. Ας πάρουμε τον τομέα του γάλακτος. Οι τιμές υπαγορεύονται όχι τόσο πολύ από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους προμηθευτές, αλλά από την αγοραστική ισχύ των ε, αυτών που αγοράζουν από τους προμηθευτές. Ε, για τις τηλεπικοινωνίες το ίδιο ισχύει. Μήπως έχουμε ε, βρεθεί σε μια κατάσταση όπου έχουμε ε, ανταγωνισμό. Γιατί το λέω αυτό. Όταν οι οικονομικοί φορείς παίρνουν την άδεια ε, υπάρχει αδιαφάνεια ως προς τις πρακτικές τους. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες καταπολέμησης του φαινομένου, αλλά δεν είμαστε πεπισμένοι ότι είναι υγιής η κατάσταση στην αγορά. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ε, ε, σε μεγάλο βαθμό υπήρξε κρατική παρέμβαση αλλά πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να εξετάσουμε το αν αυτές οι παρεμβάσεις οδήγησαν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Μακροπρόθεσμα, αυτό πρέπει να μας απασχολήσει τι είναι. Είδαμε ότι ε, έχουμε διάφορους θεσμούς βάσει της αρχής του too big to fail, ότι παρά είναι μεγάλες για να αποτύχουν και χρειάστηκε να διασώσουμε αυτούς τους θεσμικούς φορείς αλλά μήπως τώρα δημιουργούμε πάλι έτσι μεγάλους θεσμούς. Εγώ δεν έρχομαι από αυτό τον κλάδο από μια επιχείρηση έρχομαι που απασχολεί 400.000 Μήπως ε, όταν είναι μικρή μια επιχείρηση δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και όταν είναι μεγάλη, ναι μεν υπάρχει ο συστημικός κίνδυνος αλλά υπάρχει και η έλλειψη ε, αποτελεσματικότητας που οφείλεται ακριβώς στο μεγάλο μέγεθος της επιχείρησης. Ανάλογα με τον κλάδο πρέπει να δούμε ποιο είναι το ενδεδειγμένο μέγεθος των επιχειρήσεων για να μην στρεβλώνουν την αγορά, να είναι αποτελεσματικές και για να μην χρειάζεται να ε, σώζουμε εμείς αυτούς τους μεγάλους παίκτες της αγοράς όταν προκύπτει η ανάγκη. Τώρα άλλες δύο παρατηρήσεις για να απαντήσω σε ε, κάποια πράγματα που ακούσαμε για τις κρατικές ενισχύσεις. Δεν είμαστε και πολύ υπέρ των ε, κρατικών ενισχύσεων. Μπορούν να είναι αιτιολογημένες ή όχι, ανάλογα με την περίπτωση στις αναδυόμενες βιομηχανίες που πρέπει να βοηθήσουμε σε αρχική φάση μπορεί να χρειάζονται. Για το Airbus παραδείγματο χάρη πότε δεν θα είχε μεγάλη επιτυχία στην αεροδοστιακό τομέα αν δεν είχε αρχικά κρατικές ενισχύσεις. Δεν λέω ότι συνεχίζει να χρειάζεται τέτοιες ενισχύσεις ε, η Airbus αλλά δεν θα ήταν παγκόσμιος παίκτη αν δεν είχε λάβει αρχικά αυτές τις ενισχύσεις. Και οι σε μεγάλη κλίμακα προσφεύγουν σε αυτές τις ε, κρατικές ενισχύσεις. Δεν θέμα καλού και κακού εδώ. Ε, τώρα στις πράσινες τεχνολογίες και αναδυόμενες βιομηχανίες χρειαζόμαστε άμεσες ενισχύσεις, όχι ε, κρατικές ενισχύσεις, όχι άμεσες, αλλά φορολογικά κίνητρα, μέχρι ότου να διαμορφωθεί η αγορά. Και μόλις διαμορφωθεί μετά μπορεί να πετάξει με τα δικά του φτερά και να κόψουμε εμείς τις ενισχύσεις. Μπορούμε να μιλάμε για στρατηγικές εξόδου και από αυτή την πλευρά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να καταργήσουμε σταδιακά τις κρατικές ενισχύσεις. Είναι θέμα χρονισμού. Χρειαζόμαστε κρατικές ενισχύσεις επίσης ε, για να μην έχουμε ένα ε, σοβαρό σεισμό όπως αυτός που σημειώθηκε στις χρηματοπιστωτικές αγορές ε, για να μην επαναληφθεί αυτό πρέπει να προσέξουμε πώς θα αποσύρουμε τις κρατικές ενισχύσεις δηλαδή θα σκάψουμε το λάκκο μας αν θα αποσύρουμε υπερβολικά γρήγορα θα θέλαμε να, όμως να αντί, αντίθετα να επιστραφούν κρατικές ενισχύσεις που αντιβαίνουν στις κοινοτικέ πολιτικές. Παραδείγματο χάρη για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών υπάρχει πολύ σοβαρή πολιτική και ξέρουμε ότι υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις που αντίκεινται σε αυτή την πολιτική και το γνωρίζουμε. Βέβαια θα μου πείτε ότι αυτό δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, αλλά πιστεύω ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατό να αποσυρθούν αυτές οι ενισχύσεις, διότι πλήττουν ε, είναι επιζήμιες ε, για τις προσπάθειές μας να προωθήσουμε την πράσινη οικονομία. Αυτά για τις κρατικές ενισχύσεις. Ε, δεύτερον, για τα πρόστιμα. Όταν υπάρχει η παραβίαση της πολιτικής ανταγωνισμού, θέλουμε πρόστιμα χρηματικές ποινές ανάλογες προς το οικονομικό πλεονέκτημα που έχει κάποιος αν δεν σεβαστεί την νομοθεσία. Εάν παραβιάσει η επιχείρηση με την νομοθεσία και πληρώσει το πρόστιμο αλλά παρόλα αυτά βγάλει λεφτά, ε, είναι κίνητρο για να συνεχίσει ε, να παραβιάζει την νομοθεσία αυτή η επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι αν εισέλθουν σε ένα ολιγοπόλιο αν ε, διαφύγουν από το νομικό πλαίσιο ε, θα πρέπει να νιώθουν ότι διατρέχουν τον κίνδυνο να αφανιστούν. Αυτό πρέπει να καταφέρουμε. Ευχαριστούμε. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτ. Ο κύριος Φέρμπερ έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα μόνο να κάνω κάποιες παρατηρήσεις από τις αρχές γιατί πιστεύω ότι το έτος 2008 βεβαίως ε, ήταν πολύ σημαντικό στην πολιτική ε, ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κατέδειξαν αυτό άλλωστε και οι τοποθετήσεις των συναδέλφων. Έχουμε την αντικειμενική εφαρμογή ε, των συμπεφωνημένων κανόνων και την πραγματικότητα στην οικονομία που αποκλίνει από τους κανόνες. Και όταν η κατάσταση είναι έκτακτη θα πρέπει να προσαρμόζονται ή να ερμηνεύονται διαφορετικά οι κανόνες του παιχνιδιού ενδεχομένως. Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολη και συναρπαστική όμως υπόθεση, γιατί τίθεται τα θεμέλια για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον με πολλά θέματα. Να θυμίσω ξανά αυτό. Στη συνέχεια, Έχουμε διάφορους κανονισμούς ε, που τα επόμενα χρόνια θα αναθεωρηθούν και θα ήθελα το Κοινοβούλιο να πάρει θέση σαφή και ξεκάθαρη. Πρέπει να πω ότι ενοχλήθηκα που για τις ασφάλειες κάναμε επιστολή και μόνο. Η δική μου ομάδα ήθελε να αναβληθεί, ήθελε να αλλάξει η κατάσταση, αλλά στην αρχή της παρούς θητείας, από ό,τι φαίνεται, είχαμε πιο σημαντικά θέματα να ασχοληθούμε παρά με αυτούς τους κανονισμούς ε, για τις επιχειρήσεις. Ε, πρέπει να ασχοληθούμε πιο σοβαρά με αυτά τα θέματα αυτά, γιατί μετά από 50 χρόνια πολιτικής ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, θα πρέπει να σκεφτούμε τώρα τι θα γίνει στο μέλλον μετά τη θέση σε ισχύ της τη Λισαβόνας και να περάσουμε και σε ένα εκδημοκρατισμό στην επιβολή των κανόνων του παιχνιδιού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως ε, ρόλο την εφαρμογή και την υλοποίηση και το σεβασμό γιατί είναι εκτελεστικό όργανο. Δεν μπορεί όμως το εκτελεστικό όργανο να αποφασίζει και να κοινοποιεί την απόφασή του στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, και καλό θα ήταν το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει και την έκθεση αυτή τη κυρία Σινετφέλτ για να δούμε τι γίνεται με τι αποφάσει του Συμβουλίου τη δεκαετία του 60, α πούμε, Μήπως είναι επαρχιωμένες ισχύουν ακόμα, συνάδουν με αυτά που πετύχαμε πλέον με τη συνθήκη της Λισαβόνα. Επαναλαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει να αναμειχθώ στη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς εφαρμόζονται οι κανόνες. Καθόλου. Αυτό που θέλω είναι να παίζει και το Κοινοβούλιο όμως ε, στη χάραξη των κανόνων. Διότι η αλήθεια είναι ότι κάθε χώρα έχει τα προβλήματά της, ακούστηκαν πολλά τι κάνουμε με τις μικρομεσαίες, τι κάνουμε με τις ε, ε, δημοτικές ενισχύσεις της τοπικές αυτοδιοίκησης για παράδειγμα, γιατί στη δική μου περιφέρεια έχουμε εμεί δήμους και κοινότητες με ίδιο προπολογισμό που ενισχύουν τις επιχειρήσεις. Τι γίνεται σε σχέση λοιπόν με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό ή όχι. Ε, τι γίνεται με τις οριακές περιπτώσεις, δεν απλουστεύουμε αυτά τα πράγματα και αν δεν έχουμε συνέπεια και συνέχεια και έχουμε μεμονωμένες αποφάσεις αναπερίπτωση για να διορθώνουμε αυτά επιμέρους δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί αυτός που ελέγχει και εκτελεί ε, μία απόφαση να τη λαμβάνει κιόλα. Λοιπόν, να συζητήσουμε τι γίνεται με τη συνδίκη τη τι συνέπειες έχει και ποιος θα ορίζει κανόνες κανόνε του παιχνιδιού για να τους ελέγχει στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Και όλα αυτά θα τα κάνουμε με ένα νέο, μια νέα επίτροπο που ελπίζουμε προσεχώς να έχουμε πιστεύω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη κοινοβουλευτική διάσταση όλη αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Φέρμπερ. Θα μιλήσω κι εγώ πριν κλείσουμε τον κατάλογο με την τοποθέτηση της κυρίας Μπερές που μόλις ζήτησε το λόγο. Συμφωνούμε όλοι ότι ζήσαμε μία περίοδο πάρα πολύ ε, επίμαχη. Σε καιρούς πολέμου ε, επιβλήθηκε το δίκαιο του πολέμου, δηλαδή ε, ανιστάλησαν όλα όσα ισχύουν σε καιρό ειρήνης. Γίνεται ε, λόγω στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διάφορες ανακοινώσεις. Ε, δύο ανακοινώσεις έγιναν για τα χρηματοπιστωτικά και ένα για την πραγματική οικονομία. Η δεδηλωμένη πρόθεση και στόχο αυτών των ανακοινώσεων, όπω άλλωστε ομολογεί για το κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να εξασφαλιστεί ουδετερότητα ή η ισότητα μεταξύ των διαφόρων φορέων τη αγορά. Να αποτραπεί οποιαδήποτε εμφάνιση στρέβλωση ανταγωνισμού στην αγορά και είπαμε ότι οι διατάξει αυτέ είναι πάντα προσωρινέ και δεν θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα πιο διαρθρωτικά ή πιο οριστικά θα ήταν καλό λοιπόν η συγγήτρια στην έκθεσή της να διευκρινίσει αν οι στόχοι αυτοί ε, πληρώθηκαν, δηλαδή εάν αυτό που είχε δηλώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είχε στόχο, το πέτυχε ένα αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Αναλύουμε τα διάφορα στοιχεία της στρατηγικής εξόδου από την κρίση για να επανέλθουμε στην ομαλότητα και ε, στους κανονισμούς που ισχύουν σε κανονικές περιόδους. Λοιπόν, θα ήταν ε, χρήσιμο να μάθουμε τι γίνεται από τα μεταβατικά μέτρα και τα προσωρινά μέτρα. Αποκομίσαμε μόνιμα πλεονεκτήματα και διαρκή. Παράδειγμα, κάποιες τράπεζες έκαναν αύξηση κεφαλαίου με κρατικές ενισχύσεις ή για την τόνωση της ρευστότητας και του ενεργητικού τους. Δεν θα είχε πολύ μεγάλο νόημα οι τράπεζες αυτές τώρα να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα τη στιγμή που αναλύουμε το επίπεδο κεφαλαίου των διαφόρων τραπεζών στις διάφορες οδηγίες που έχουμε για το θέμα αυτό. Γιατί δεν θα ήταν και πάρα πολύ ισότιμο, έτσι. Δηλαδή κάποιες τράπεζες που ενισχύονται από τα κράτη για να τονωθεί η λειτουργία τους έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες. Κάποια στιγμή πρέπει να τερματίζονται οι, οι, οι κρατικές ενισχύσεις. Και για τα υπόλοιπα λίγο έχω να πω. Δίνω μόνο το λόγο στην κυρία Περβάς Μπερές και μετά και στην ε, κυρία Χιούμπνερ που μου το ζήτησε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαίρω την εισηγήτρια για τη στάση την οποία επιλέγει. Έχουμε να κάνουμε με μια επαναλαμβανόμενη προσπάθεια όπως και άλλες αιτήσιες πάση περιπτώσει εκθέσεις προσπάθειες που κάνουμε έτσι και η έκθεση για τον ανταγωνισμό στην ουσία είναι μια προσπάθεια να επαληθεύσουμε το σεβασμό των νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν γίνει δεκτές στο παρελθόν. Θα θέσω λοιπόν τρία συγκεκριμένα θέματα. Θα ξεκινήσω από το πιο συγκεκριμένο για να καταλήξω στο πιο γενικό. Αυτό το πιο συγκεκριμένο είναι κάτι το οποίο απασχολεί όχι μόνο εμένα, είναι το θέμα του ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Το έχουμε κάνει και πέρυσι και πρόπερσι για την περίπτωση των σταζιέρ, για την περίπτωση των στάζ. Αυτές είναι πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ σε πολύ μεγάλες ιδιαίτερα επιχειρήσεις και πίσω από τον πολλαπλασιασμό των στάζ, ιδιαίτερα προς τους νεοτέρους, έχει υπάρξει μια σαφέστατη χειροτέρευση των συνθήκων εργασίας και σε επίπεδο ανταγωνισμού υπάρχει κάτι το οποίο μας επιτρέπει να μπούμε στη συζήτηση για να δούμε ακριβώς πώς μια επιχείρηση μέσω του πολλαπλασιασμού των θέσεων σταζιέρ στην ουσία χρησιμοποιεί ένα πλεονέκτημα ανταγωνιστικό. Αυτά για τα στάζ. Το δεύτερο θέμα, το οποίο θα έλεγα δεν πρέπει να αγνοήσουμε στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης, είναι οι μεγάλες εταιρείες και οι, μεγάλες, οι μεγάλοι ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων. Νομίζω ότι και εδώ θα συμφωνήσω με την εισηγήτρια. Το τρίτο θέμα είναι λίγο πιο γενικό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε επίση συζητήσει στο παρελθόν, το της εντολής δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν βλέπουμε ότι χρησιμοποιούμε ένα ορισμό της πολιτικής ανταγωνισμού που εν πολλής αγνοεί πραγματικότητες οι οποίες είναι αντίθετες με, τις, με τους κανόνες τους βασικούς του ανταγωνισμού. Και μιλάω για τις εταιρείες αξιολόγησης, για τις μεγάλες εταιρείες ελέγχου των λογιστικών των εταιριών και για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο είναι αντίθετο όχι μόνο με το γράμμα της συνθήκης αλλά σίγουρα με το πνεύμα της συνθήκης. Νομίζω ότι μια σωστή πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση να γίνει σεβαστή έτσι ώστε οι χώρες μας να μην διατρέχουν κίνδυνου στον τομέα αυτό αδικαιολόγητα. Εν πάση περιπτώσει η έκθεσή σας θα είναι πολύ χρήσιμη για να κατανοήσουμε και το τι συνέβη το 2008. Ξέρουμε ότι δεν έχουν εφαρμοστεί όλα τα μέτρα τα οποία είχαμε ζητήσει για το 2008 και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα η Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό και η Επίτροπος εφάρμοσαν τους κανόνες στην περίπτωση έγκρισης των προγραμμάτων υποστήριξης προς τα πιστοτικά ιδρύματα. Τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοιτάξτε εδώ έχει ξεσπάσει πυρκαγιά δεν θα πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα μίζεροι σε σχέση με τη χορήγηση της βοήθειας. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό όταν αργότερα δούμε το τι αποκατάσταση των προβλημάτων έχει υπάρξει. Και τελικά θα μας πούνε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή τώρα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, για τον οποίο να δούμε οι τράπεζες ε, έχουν ενισχύσει τη θέση τους και μάλιστα ορισμένες υπερβολικά στις αγορές. Ίσως να με κατηγορήσετε για ουτοπίστρια, αλλά μια σωστή πολιτική ανταγωνισμού θέτει σαφώς ε, και λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κανόνων. Δεν το ζήτησε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν εξετάζει μόνο εκ των υστέρων τα αποτελέσματα μιας προσπάθειας αποκατάστασης μιας επιχείρησης, στην ουσία λειτουργεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της αν έπρεπε εξ αρχής ε, να θέσουν προϋποθέσεις, τότε θα έπρεπε να διαπραγματευτούν με τα κράτη-μέλη, τότε θα έμπαιναν σε μια διαδικασία η οποία δεν θα είχε τέλος. Έχει λοιπόν ακολουθηθεί από την Κομισιόν μια διαδικασία η οποία ναι μεν στάθηκε σε μια πρώτη φάση χρήσιμη για την εσωτερική αγορά, για μια αποκατάσταση της υγείας θα έλεγα της, ε, του πιστοτικού τομέα, του τραπεζικού ε, τομέα ε, ενώ από την άλλη θέματα τα οποία θα έπρεπε να είναι προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος αυτού όπως το θέμα των αμοιβών των στελεχών, το θέμα της ενίσχυσης δανειοδοτικά από τα πιστοτικά ειδήματα των μικρομεσαίων κτλ. δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ε, για να κλείσει τη συζήτηση αυτή η κυρία Χιούμπνερ. Ίσως ε, να μην φάνηκε ότι ήθελα να μιλήσω προηγουμένως, αλλά θα ήθελα το λόγο, γιατί έχω την αίσθηση ότι η έκθεση αυτή είναι μια πολύ σημαντική έκθεση. Δεν είναι μια έκθεση τύπου business as usual. Οι καιροί είναι καιροί γεμάτοι προκλήσεις, είναι καιροί που δημιουργούν κινδύνους και θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα. Να αναφερθώ σε δύο από τα θέματα στα οποία ήδη αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι και που συνδέονται με τις κρατικές βοήθειες. Ξέρετε ότι δόθηκαν μαζικές στηρίξεις από πλευράς των κρατικών προϋπολογισμών και αυτό το ζήτησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρχή του χρόνου. Ήταν τα, τα λεγόμενα μέτρα διάσωσης κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων Υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες βέβαια για τέτοιου είδους προγράμματα στήριξης για την ολοκλήρωσή τους εννοώ. Και υπάρχει κι άλλο ένα θέμα το οποίο επιβαρύνει αυτού του είδους τα μέτρα, ότι τα ωφέλη τα οποία δόθηκαν κυρίως στις τράπεζες έπρεπε να περάσουν στην πραγματική οικονομία. Και γι' αυτό σήμερα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα φορά να μην λειτουργήσουν με διαφορετικό τρόπο γιατί αυτό θα ήταν σοβαρό λάθος. Αυτό το οποίο πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι βασικά δύο πράγματα, δύο ανηλυμένες υποχρεώσεις. Πρώτον, να μας πούν πώς ακριβώς έχουν προοδεύσει αυτές οι διαδικασίες βοήθειας προς συγκεκριμένα τμήματα της οικονομικής δραστηριότητας και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει μια ανάλυση σχετικά με το αν τα κέρδη στα οποία έχουν περάσει πλέον πολλές από τις επιχειρήσεις που βοηθήθηκαν από τον κρατικό κορβανά έχουν βοηθήσει την πραγματική οικονομία. Η Επιτροπή θα ήθελε το λόγο. Σύντομα, Πρόεδρε. Δεν θα σχολιάσω τα μεμονωμένα θέματα τα οποία έθεσαν πολλοί από τους συναδέλφους σας. Θα σχολιάσω όμως την βασική γραμμή την οποία ακολουθεί η συγχύτρια. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή πράγματι προσπαθεί να παρουσιάσει την πραγματικότητα με συγκεκριμένο συνεκτικό τρόπο και δεν αγνοεί τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον προηγούμενο χρόνο για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση. Έχουμε εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα, έχουμε εφαρμόσει συγκεκριμένους κανόνες, έχουμε βοηθήσει τις αναδιαφρώσεις των πιστοτικών ε, ε, οργανισμών για να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητά τους όπως επίσης και τον υγιή ανταγωνισμό. Θα θέλαμε να συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας για το πώς θα αντιδράσουμε στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσής μας στα σχόλια τα οποία κάνει το Κοινοβούλιο. Στο παρελθόν δεν αντιδράσαμε πάντα με τον κατάλληλο τρόπο στα σχόλιά σας ε, και πρέπει να σας δώσουμε εξηγήσεις γιατί κάποιες από τις προτάσεις σας τις κάναμε δεκτές ενώ κάποιες άλλες όχι. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας δώσουμε όλες αυτές τις εξηγήσεις. Θα ήθελε να κλείσει η συζήτηση η συγγήτρια παρακαλώ. Κάποιοι είπαν ότι ίσω είναι υπερβολικά φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα, αλλά ακούγοντα του συναδέλφου, βλέπω ότι υπάρχει ομοθυμία σε μεγάλο βαθμό και μπορεί να μην χρειαστεί καν η προθεσμία που έχουμε θέσει. Νομίζω ότι συμφωνούμε για διάφορα στήματα με τους συναδέλφους. Πρώτον, σχετικά με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σχετικά με τη διαδικασία λήψη πολιτικών αποφάσεων, Συμφωνώ με τον κύριο Φέρμπερ για αυτό το θέμα και μέσα στην έκθεση θα τονίσουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου να είναι υπόλογη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ταυτόχρονα θα ήθελα να πω το εξής ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ούτω ώστε να μην εκτεθεί σε εθνικές πολιτικές πιέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντική και σίγουρα βέβαια θα καταφέρουμε να βρούμε μια ισορροπία. Δεύτερο σημαντικότατο ζήτημα, οι κρατικές ενισχύσεις. Και βλέπω ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχει συνένεση. Ο κύριος Μπούλμαν ε, έθεσε το ε, δάχτυλο επί του τύπου των ήλων μιλώντας για τη δυνατότητα παρέμβασης η όλη διαδικασία όμως θα πρέπει να έχει ως στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας κρατικής ενίσχυσης Επίσης, να διαπιστώσουμε αν εκπληρώθηκαν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Δεν μιλώ μόνο για την οικονομική ανάκαμψη, γιατί υπάρχουν και επιπρόσθετοι ε, στόχοι. Η πράσινη ανάκαμψη, ε, η χάρη του να περάσουν τα πλεονεκτήματα των κρατικών ενισχύσεων στην πραγματική οικονομία και να διαπιστώσουμε αν εκπληρώθηκαν, ξαναλέω, επιδιωκόμενοι στόχοι. Είναι συμφωνώ με τον ε, κύριο Μπούλμαν ότι αυτό είναι ο ρόλο των εθνικών αρχών ε, σε περιπτώσει κρίση να παρεμβαίνουν, αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν πρόκειται για μάνα εξ ουρανού. Ταυτόχρονα έχουμε αυξανόμενα δημόσια χρέη και θα χρειαστούν χρόνια ή και δεκαετίες ε, για να ξαναμπούμε στο σωστό δρόμο, μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και άρα δεν θα έχουμε αρκετά κονδύλια για πράγματα που μας ενδιαφέρουν, η παιδεία, το περιβάλλον, ε, η, επένδυση πράσινες τεχνολογίες όπως μας είπατε, η υγειονομική περίθαλψη, πράγματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Κάθε σέντ που δίνουμε για κρατική ενίσχυση ε, πρέπει να δαπανάτε συνετά και έχουμε ευθύνη να ελέγχουμε ε, αν όλα αυτά ισχύουν και επίσης να είναι και υπόλογοι, ξαναλέω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την νομοθεσία αντιτράς και τις συγχωνεύσεις ε, δεν συζητήθηκε πολύ αυτό το θέμα αλλά από τα λίγα που άκουσα νομίζω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε συμφωνία Και έχοντας ακούσει τους συναδέλφους ε, θα πρότεινα και συντομότερη προθεσμία. Το αργότερο το Μάρτιο θα ήθελα να εγκριθεί η έκθεση γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και μεγαλύτερη επιρροή. Θα προετοιμάσω λοιπόν το Σαββατοκύριακο το σχέδιο, θα το στείλω για μετάφραση την ερχόμενη εβδομάδα. Θα το στείλω στους και στα αγγλικά και το ταχύτερο δυνατό θα προσπαθήσω να κλείσω το θέμα. Α, ναι. Και μην το ξεχάσω, ήθελα να σας πω, ο κύριος Σουβάπ νομίζω δικαίως ανέφερε το ότι θα πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων κάποιες μορφής. Ε, δεν χρειάζεται ε, κανονική ακρόαση νομίζω γιατί μας τρώει πάρα πολύ χρόνο από τις τακτικές συνεδριάσεις μας αλλά ίσως ε, μια συνεδρία συντονιστών ανοιχτή κάποια, κάποιας μορφής συνεδρίασης εμπειρογνωμών και θα βρούμε ποιους εμπειρογνώμους θα καλέσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Σοφή. Οκρώνεται εδώ η συζήτηση για το σημείο αυτό. Για την έκθεση της πολιτικής ανταγωνισμού 2008. Μικρή διακοπή για τρία λεπτά για να πάει η ώρα και τέταρτο ακριβώς για να αρχίσουμε την ψηφοφορία όπως είχαμε ε, προβλέψει στην ημερήσια διάταξη. Um, λοιπόν, έχουμε ψηφοφορίες, ξέρετε. Μία ψηφοφορία και σύντομη, ελπίζω. got their voting Έχετε όλοι τους καταλόγους ε, για την ψηφοφορία. Το μικρόφωνο μου είναι ανοιχτό και δουλεύει, δεν με ακούτε. Βάλτε τότε κανένα ακουστικό. Λοιπόν, είστε έτοιμοι όλοι να ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε την έκθεση λοιπόν του κυρίου Μπούλμαν. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας. Ελπίζω να είναι και σωστή η λίστα που έχω. Τροπολογία 5 πρώτη. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμό 12 του κυρίου Σμιτ έχει αποσυρθεί και θα περάσουμε στη συμβιβαστική α. Ψήφι πέρα παρακαλώ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Α, τώρα τι έχουμε. Sorry, Amendment 7, recital 8. Yeah, that's right. Amendment, uh, that, that, that, that, all... Ah, μάλιστα. Οι υπόλοιπε τη ενότητα αυτή καταπίπτουν και περνάμε στην τροπολογία περθών 7 ψήφι υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. Η τροπολογία περθών 1 ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται που σημαίνει ότι 8 καταπίπτει 2 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται που σημαίνει ότι καταπίπτει 10 και πάμε στην τροπολογία 11 γιατί η 3 έχει υποσυρθεί Α, έχει καταπέσει, λέει ο συντάκτη ο κύριο Φέρβερ, ωραία. Οπότε... Έχουμε την 4 του εισηγητή ψηφιπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται επίση. Μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα, σα παρακαλώ. Κάντε λίγη σχέση σας παρακαλώ. Το κείμενο όπω τροποποιήθηκε Ψήφιπε Against. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται προφανώς. Και το νομοθετικό ψήφισμα, Ψήφιπε Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Okay, Λοιπόν, προχωρούμε στη δημόσια ακρόαση. Είμαι βέβαιη ότι θα αφιερώσουμε όλο το χρόνο σε αυτή την ακρόαση. Αρχίζω ένα-δύο λεπτά νωρίτερα για να τελειώσουμε με τα διαδικαστικά, με τις συστάσεις και τα λοιπά, για να περάσουμε στην ουσία πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, βλέπω ότι το διασκεδάζεται και πίσω όλα θα πρέπει να αρχίσει η ακρόασή μας. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μέχρι τις 10.30. Λοιπόν, να σας πω πώς θα προχωρήσουμε το κείμενο που περιλαμβάνει τα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών το έχετε λάβει είναι όλοι εξέχουσε προσωπικότητες και πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Δεν θα αναρωθώ στην παρουσίαση του καθενός για να τους δώσω ε, το χρόνο να μιλήσουν. Δεν θα τους εκθιάσω από πόσο καλοί και σπουδαίοι είναι. Ζητώ συγγνώμη αν φανεί αυτό αγενές. Έχετε τα στοιχεία στα χέρια σας για να καταλάβετε περί ποιων ανθρώπων ε, πρόκειται. Αν δεν τους βλέπετε που κάθονται, κάθονται από την τέταρτη σειρά και πίσω στη μέση περίπου. Στο μεσαίο διάζωμα για να το πω έτσι. Μετά την εισαγωγή μου θα δώσω σύντομα το λόγο στον εισηγητή μας, τον Ζαν Πολ Γκοζές, που θα πει μερικά λόγια και μετά Θα έχουμε μία ώρα για να ακούσουμε τους ομιλητές, τους εμπειρογνώμονες και θα τους παρακαλέσω όλους να τηρήσουν το χρόνο που τους έχει δοθεί. Επίσης πρέπει να σας πω ότι θα σας στείλουμε ηλεκτρονικά τα έγγραφα με τις παρουσιάσεις των ομιλητών μας μετά τη συνεδρίαση. Και όπως ακούσαμε προηγουμένως ο κύριος Ρενέ Χόφμαν, αναπληρωτής ε, γραμματέας του CTUC θα μιλήσει με την κυρία Τζάνετ Βίλιαμσον ε, που είναι και εκείνη από την Ευρωπαϊκή ε, Ομοσπονδία Συνδικάτων. Και βεβαίως ως ήθιστε μεταδίδεται απευθείας και στο διαδίκτυο η συνεδρίαση. Το Κοινοβούλιο ζήτησε μελέτη αντικτύπου η οποία έχει φτάσει. Η πρώτη έχει δημοσιευθεί και η δεύτερη αναμένεται περί τα τέλη του μηνός ε, Νοεμβρίου. Δεν νομίζω χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω για τα διαδικαστικά και την πορεία της ακρόασης. Ε, με χαρά δίνω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ζανπόλ Γκοζές, για να μας πει και εκείνο ε, μερικά εισαγωγικά λόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι οι προσωπικότητες τις οποίες έχουμε καλέσει να μπορέσουν να εκφραστούν πάνω σε ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα, ένα θέμα περίπλοκο. Περίπλοκο γιατί το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας είναι ευρύτατο καλύπτει ότι δεν έχει σχέση με την προηγούμενη οδηγία και διακυβεύονται πάρα πολλά συμφέροντα, συμφέροντα μερικές φορές θα έλεγα αντιτιθέμενα μεταξύ τους. Ένας από τους συνεισηγητές μου είπε ότι έχουν παρέμβει πάρα πολλά λόμπι, ένας πολύ μεγάλος αριθμός λόμπι έχουν πιέσει ιδιαίτερα. Εγώ συνεχίζω να ε, συναντώ αυτούς οι οποίοι μου ζητούν συναντήσεις και έχω κλείσει τον χρόνο μου μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009. Έχω χρόνο για την επόμενη χρονιά. Αυτό το οποίο περιμένουμε λοιπόν από την ακρόαση αυτή και το workshop που θα ακολουθήσει το απόγευμα είναι κάποιες παρατηρήσεις πάρα πολύ συγκεκριμένες. Ο εισηγητής δεν γνωρίζει τα πάντα, δεν είναι σοφός. Αυτό το οποίο προσπαθεί είναι επί τη βάση των εμπειριών τις οποίες έχει συλλέξει, επί τη βάση των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του, να ρυθμίσει κάποιες ε, νομοθετικές θα έλεγα, ε, νομοθετικό επίπεδο ρυθμίσεις, οι οποίες να είναι απλές, συγκεκριμένες, κατανοητές, να ανταποκρίνονται ε, στα συμφέροντα των πολιτών και όλων των εμπλεκομένων μεταξύ των οποίων και τη βιομηχανία. Πολλοί έρχονται και μου λένε ότι η οδηγία καλή είναι, αλλά ξαφνικά αρχίζουν να την απεκδίουν θα έλεγα και την αφήνουν στο τέλος γυμνή και ανυπεράσπιστη. Τέτοιου είδους λογικές δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο η οποία λέει ότι ε, στα πλαίσια της κρίσης και ακόμα και αν τα hedge funds, τα εναλλακτικά αυτά funds δεν είναι η βασική αιτία της κρίσης, παρόλα αυτά ε, δεν θα πρέπει να υπεκφύγουν ρύθμισης και ελέγχου εποπτείας, θα πρέπει να είναι όσο πιο αποτελεσματική γίνεται αυτή η εποπτεία και γι' αυτό θα σας ακούσουμε στις παρατηρήσεις που θα κάνετε και στην περιγραφή των αρμοδιοτήτων σας και των εμπειριών σας. Thank you very much. Um, Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περιθώριο χρόνου. Οι πρώτες παρουσιάσεις είναι εξ ονόματος της ΙΟΣΚΟ και της ΣΥΖΑ. Ε, πρώτη Βερένα Ρος, συμπρόεδρος της ομάδας ε, κρούσης για την έκθεση Hedge Funds Oversight της ΙΟΣΚΟ, που είναι διεθνής οργανισμός ε, των επιτροπών για τις securities. Η Βερένα φαίνεται έτοιμη να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι που με προσκαλέσατε σήμερα στην Ακρόαση. Βερίνα Ρος ε, λέγομαι ε, και είμαι πρόεδρος ε, στην Task Force της ΙΟΣΚΟ για τις χρηματοπιστωτικές ενότητες, της μη ρυθμισμένες της ΙΟΣΚΟ. Ε, και εκπονούμε, εκπονήσαμε νωρίτερα φέτος ε, την έκθεση για την εποπτεία για τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, τα hedge funds. Μετά από αίτηση της μας ζητήθηκε να εξετάσουμε την κατάσταση για τις μη ρυθμισμένες χρηματοπιστωτικές ενότητες. Δεδομένου του ενδιαφέροντας της G20 για αυτά τα ταμεία, η Task Force μας αποφάσισε να εστιάσει τις εργασίες της στα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και ε, να μην ασχοληθεί με άλλες ε, μονάδες ε, όπως παραδείγματο χάρη τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια γιατί μας έχουν απασχολήσει στο παρελθόν. Στην τελική έκθεσή μας ε, που εκπονήθηκε τον Ιούνιο αναφέρουμε ότι πολλές παρατηρήσεις και πολλά συμπεράσματα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους συμμετέχοντες της αγοράς. Σε άλλες μονάδες που κατέχουν ή ελέγχουν μεγάλες μονάδες ιδιωτικών κεφαλαίων η διάκριση ανάμεσα στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου είναι σημαντική όταν περάσουμε στις λεπτομέρειες ε, των προτάσεων που εποβάλλουμε. Καταρχάς να τονίσω ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στους γενικούς στόχους ρύθμισης της ΑΕΟΣΚΟ για το χρηματοπιστωτικό τομέα και των στόχων της ε, οδηγίας. Πρώτα απ' όλα, ε, η προετοιμασία της οδηγίας και η έκθεση της ε, ΙΟΣΚΟ είναι απαντήσεις που δίνουμε σε προβλήματα που προέκυψαν από την χρηματοπιστωτική κρίση και ε, προέρχονται από τη δέσμευση που έχουν λάβει αρχηγικά των κυβερνησιών στην G20 για να βελτιώσουν την εποπτεία όλων των παικτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές όταν υπάρχει συστημητικός κίνδυνος για ολόκληρη την αγορά ή τμήματά της. Πιστεύω ότι και οι κοινοτικές αρχές και η ΙΟΣΚΟ αναγνωρίζουν ότι η έσχατη χρηματοπιστωτική κρίση δεν προκλήθηκε από τα hedge funds. Στην έκθεση που δημοσιεύσαμε το Μάρτιο του 2009 το αναφέραμε αυτό με πυγμή και αναγνωρίσαμε παρόλα αυτά ότι οι δραστηριότητε των ταμείων αντιστάθμισης κινδύνου μπορούν να οξύνουν ε, τι επιπτώσει τη κρίση. Ε, Παραδείγματο χάρη διότι τα hedge funds μα με άλλου συμμετέχοντε τη αγορά ε, πρέπει οπωσδήποτε να μειώσουν την έκθεσή του λόγω των περιορισμών ρευστότητα, ε, γιατί οι επενδυτέ, παραδείγματο χάρη, σε μεγάλο βαθμό εξόφληση των κινητών αξιών του. Ε, και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα hedge funds στι χρηματοπιστωτικέ ε, αγορέ πρέπει να αντιμετωπιστούν από μια γενική ρυθμιστική δραστηριότητα. Άλλα κοινά στοιχεία είναι ότι και στη ΙΟΣΚΟ και η Οδηγία να γνωρίζουν την ανάγκη που υπάρχει για την καταγραφή και την αδειοδότηση των διαχειριστών των επενδυτικών ταμείων χρειάζονται διεθνή πρότυπα για την καταχώρηση καθώς και για την ε, εποπτεία αυτών. Επίσης χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια για τους ίδιους τους επενδυτές, να ε, ε, συμμόρφωση με τους κανόνες για την κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού και σχετικά με την απόδοση των επενδυτικών ταμείων, αλλά αυτά είναι σημαντικά. Στην ΑΕΟΣΚΟ μας απασχολεί η μόχλευση, η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού, η διαχείριση του κινδύνου και επίσης η σημασία της ε, Συνεργασία των εποπτικών αρχών. Ε, βέβαια δεν έχουμε προτείνει αυστηρά όρια για τη μόχλευση, ούτε και έχουμε θέσει κεφαλοχικές ε, απαιτήσει για τους διαχειριστές των ελλακτικών επενδυτικών ταμείων. Στιάσαμε την προσοχή μας στην ανάγκη για τους ρυθμιστές να έχουν τις κατάλληλες πληροφορίες από τους διαχειριστές των επενδυτικών ταμείων, ούτως ώστε εμείς οι ρυθμιστικές αρχές να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε τους συστημικούς κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν αυτοί οι παίκτες της αγοράς. Ε, υπάρχει συνοχή ανάμεσα στην προσέγγιση που ακολουθείται στην οδηγία και στι εργασίε τη ε, ΙΟΣΚΟ και τώρα θα ασχοληθώ με τι διαφορέ ανάμεσα στα δύο. Η πιο σημαντική, κατά τη γνώμη μου, είναι η παγκόσμια διάσταση. Σε κάποιο βαθμό ξέρω ότι αυτό είναι αναπόφευκτο, διότι προφανώ ε, διαφέρουν ελαφρώ οι απόψει μα για το τι πρέπει να γίνεται στον κόσμο. Υπάρχει η διεθνή προσέγγιση και ο ορισμό των προτύπων και η ευρωπαϊκή προσέγγιση από την άλλη. Αλλά στην έκθεσή μας τονίζουμε ότι παρότι τα ρυθμιστικά πρότυπα διαφέρουν ανάλογα με το κράτος για το οποίο μιλάμε, παρόλα αυτά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οποιοδήποτε ρυθμιστικό μέτρο ή πρότυπο πρέπει να οδηγεί σε συλλογική δράση και συλλογική εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της κινητικότητας ε, του κεφαλαίου. Ε, και στη διαβούλευση που έγινε όλες οι απαντήσεις δείχνουν ότι πρέπει όντως να συγκλίνουν οι νομοθεσίες περί της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους ε, του ρυθμιστικού και για να έχουμε ισότιμου όρου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Ζακ Τελαροζιέρ νομίζω ε, κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα ότι τελικά πρέπει να έχουμε ε, ουσιαστική, ρεαλιστική ευρωπαϊκή συνεργασία προ όφελο όλων για να έχουμε μια ανοιχτή παγκόσμια αγορά. Και αυτό συνάδει με τη γνωμοδότηση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που τόνισε την ανάγκη να υπάρχει παγκόσμια συνοχή σχετικά με τα αριθμιστικά και τα υποπτικά πρότυπα. Η ανάγκη που υπάρχει για παγκόσμια πρότυπα επηρέασε τι αρχέ και προσέγγιση τη ΑΕΟσκο σχετικά με τι αρχέ και συγκεκριμένα τις ε, τελικέ συστάσεις ε, για να έχουμε σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο συμμόρφωση ε, με του όρου και τις αρχές για να αρχίσει σε παγκόσμιο επίπεδο η εποπτεία και κατά την εφαρμογή των αρχών επί των οποίων έχουμε συμφωνήσει και αυτό το κάνουμε για να μεριμνήσουμε τόσο στο μέτρο του δυνατού να έχουμε μια παγκόσμια ρυθμιστική προσέγγιση για τι διεθνεί χρηματοπιστωτικέ αγορέ που λειτουργούν αισίω. Όπω είπε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μια διεθνώ συντονισμένη δράση που θα μα βοηθήσει ούτω ώστε οι απαιτήσει να, να υπάρχει συμμόρφωση με τι απαιτήσει και από τι τρίτε χώρε, από του διαχειριστέ των εναλλακτικών επενδυτικών ταμείων, να ισχύουν δηλαδή ε, οι ίδιοι κανόνε, ούτω ώστε όσοι δεν έχουν την καταστατική του έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι το θέμα των τρίτων χωρών μα έχει απασχολήσει πάρα πολύ στα πλαίσια της ε, διαπραγμάτευσης της οδηγίας. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι μη διακριτική συμπεριφορά ως προς την προσέγγιση που ακολουθούμε είναι επωφελής ε, και για τους επενδυτές ε, και για τους καταναλωτές και για τα επενδυτικά ταμεία. Ένας άλλος ταμέας όπου πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά κοινά στοιχεία όσο θα θέλαμε ανάμεσα στις εργασίες που γίνονται από την Ιόσκο και τις εργασίες για την οδηγία είναι διαφοροποίηση των, ως προς τους διαχειριστές των εναλλακτικών επενδυτικών ταμείων. Εμείς ασχολούμαστε συγκεκριμένα με τα hedge funds ε, και όχι γενικότερα με όλα τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία και νομίζω ότι ε, θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το ε, πώς κινούνται οι σύμβουλοι, οι διαχειριστές και όλοι όσοι παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες εναλλακτικών επενδύσεων και ε, περιγράφουμε το πώς λειτουργούν τώρα τα hedge funds ε, για να δούμε ποιοι είναι ενδεχόμενοι συστημικοί κίνδυνοι και για να ε, αμβλύνουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Στο μέτρο του δυνατό, όπως σας είπα και προηγουμένως, αναγνωρίζει η ΟΣΚΟ τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα hedge funds και στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Δεν θέλουμε ένα ενίο πρότυπο για το διαχειριστή του ταμείου, γιατί δεν γίνεται λόγω της διαφορετικής φύσης των επενδυτικών ταμείων. Απλά ασχοληθήκαμε συγκεκριμένα αυτό το τμήμα της αγοράς και γι' αυτό εκπονούμε την έκθεση για αυτά συγκεκριμένα τα ταμεία. Θα κλείσω εδώ. Ελπίζω να σα εξήγησα πού υπάρχουν κοινά σημεία αλλά και διαφορέ ανάμεσα σε εργασίε που γίνονται στην ΑΙΟΣΚΟ και εργασίε που γίνονται στα πλαίσια τη οδηγία και θα επανέλθω σε αυτά τα ζητήματα να περάσουμε σε ερωταπαντήσει. Συνέχεια ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Βερένα. Αυτό δείχνει ακριβώς πόσο δύσκολο είναι να τηρήσει κανείς τον χρόνο του, διότι ε, τον υπερεύεις και είχαμε και με μία μίνι κρίση μέχρι να ετοιμάσουμε τον υπολογιστή για την επόμενη τοποθέτηση, μέχρι να διορθωθεί λοιπόν σε άφησα για μαγρικορήσεις. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Έντι Βάιμερς. Όχι. Ο εισηγητής, ο κύριος Γκοζές. Μία ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Μας μιλάτε για το χρόνο, αλλά και τα δύο εδώ έχουν σταματήσει στις 10 παρα 10 Όπω τον παλιό χρόνο που είχαμε αγροτικούς γεωργικούς μαραθωνίους που σταματούσαν το ρολόι. Καλό θα ήταν να βάλετε κανένα χρονόμετρο για να ξέρουν οι ομιλητές το χρόνο που έχουν. Ευχαριστώ. Καλώς, η Πρόεδρος. Υποθέτω ότι μπορούμε να κάνουμε το εξής. Όταν αρχίσει ο επόμενος ομιλητής και να επαναφέρουμε το χρονοδιάγραμμα. 10 και 45. Για να δούμε πόσα λεπτά θα μιλάει ο καθένα. Αλλιώ έχετε και ρολόγια. Τι το θέλει το χρονόμετρο. Λοιπόν, ο επόμενο ομιλητή είναι ο Έντι Γουάιμερ, πρόεδρο τη Caesar Δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσει. Μα λένε ότι εμεί θα αλλάζουμε τι διαφάνειε. Αν θέλετε λοιπόν να περνάτε στην επόμενη, μα το λέτε γιατί μη χειριζόμαστε εδώ το σύστημα. Ή κάντε ένα νόημα, εν πάση ε, ε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σε αυτή την τόσο σημαντική ακρόαση και βλέπω ότι είναι μεγάλη αίθουσα και σχεδόν γεμάτη. Οπότε, μάλλον είναι σημαντική ακρόαση για να έχει τόσο κόσμο. Ε, για και εγώ το χρόνο μου θα κάνω ό,τι μπορώ ε, θα ήθελα καταρχάς να αναρωτηθώ τι κάνω εγώ εδώ, δεν είναι σαφές γιατί μέχρι τώρα η Σίζαρ δεν έχει λάβει καμία θέση επί του θέματος ε, ουσιαστικά δεν συνδέεται με αυτή τη δουλειά σε επίπεδο συμβουλίου. Δεν συμμετέχουμε στο συμβούλιο και δεν μπορώ να σας παρουσιάσω καμία γνωμοδότηση εξ ονόματος της ΣΥΣΑΡ, που είναι λίγο περίεργη τώρα η θέση μου. Να έρχομαι να μιλάω για ένα θέμα για το οποίο ουσιαστικά δεν έχω ρωτηθεί και δεν έχω και ε, νομιμότητα να μιλήσω, δεν δικαιολογείται. εκτό από την προσωπική μου άποψη που είναι πιο ακαδημαϊκή και ε, όχι λειτουργική σίγουρα. Ελπίζω να καταλάβετε σε τι δινή θέση βρίσκομαι τώρα και ποιο δίλημα έχω. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας προτείνω κάποιες ιδέες ε, προσωπικές που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Δεν θα μπω Στι λεπτομέρειε έχω κάνει 27 διαφάνειες. Αν τις παρουσιάσω και 27, μέχρι τις 12 η ώρα εγώ θα μιλάω. Και δεν είναι και πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Λοιπόν, ε, οι στόχοι ε, πρώτα θα πρέπει να είναι σαφείς. Τι θέλουμε, τι επιδιώκουμε και σε τι αποσκοπούμε. Πολλά πράγματα. Πρώτον, αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου. Θα συμφωνούν όλοι ότι πρέπει να γίνει αυτό. Και ε, υπάρχει το θέμα όμως ε, της συμπεριφοράς της αγοράς. Είδαμε καταχρήσεις πρόσφατα και ξέρουμε ότι Υπάρχουν ε, κάποιοι κύκλοι ε, ανθρώπων που έχουν εσωτερική γνώση και ε, δρούν εσωτερικά. Πριν γνωρίζει το ευρύ κοινό τι γίνεται. Υπάρχει λοιπόν η σχέση του χρήστη. Του χρήστη. Τι σύστημα θα έχουμε. Το usage, το ΣΕΚΑ στα ελληνικά. Όλο αυτό το θέμα της διακυβέρνησης επίσης που δεν το έχουμε δει και ε, τα, τους κινδύνους της ε, ε χρηστής διαχείρισης ε, prudential risk. Να σας πω δύο λόγια για το πεδίο εφαρμογής. Γιατί το λέω αυτό. Έγινε στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αύριο δημοσιεύεται νέο κείμενο το οποίο μου είναι άγνωστο. Το πεδίο εφαρμογής συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Και το θέμα είναι ήταν καλή επιλογή αυτή. Νομίζω ότι το παρακάνουμε. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μερικά σημεία που βεβαίω μπορεί στο νέο σχέδιο οδηγίας να ρυθμίζονται. Οι εταιρείε ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, private holdings, είναι πολλές στην Ευρώπη. Εντάσσονται στην οδηγία ή όχι. Μετά, κάποιοι επενδυτέ, όπω επενδυτέ σε κεφάλαια κινδύνου, ε, επίση θα μπουν στην οδηγία και εκεί χρειάζεται κάποιος διαχωρισμός και ε, ε, αφενός να βγουν τα ιδιωτικά επικεντρωτικά κεφάλαια, θα επανέλθω στη συνέχεια σε αυτό, αλλά και θέματα εκτίματα αγοράς, άλλο σημαντικό και δύσκολο, ακόμα και ε, τα μία που έχουν παθητικό σε θέματα εμπορίου λοιπά Τώρα, οι θεματοφύλακες ε, depositories για τα hedge funds είναι το θέμα του usage. Είναι ένα δημόσιο εργαλείο. Δεν θα πρέπει να ε, προστατεύεται λιγότερο από τα hedge funds. Εγώ θα πρότεινα να μην βάλουμε τη ρήτρα όπως έχει σήμερα που είναι υποχρέωση αποτελέσματος αλλά να βάλουμε ένα σύστημα με πιο αυστηρούς κανόνες για τη ε, δέουσα ταχύτητα ή επιμέλεια, due diligence, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτό το καθεστώς φυλάκων, ανάλογα με τις ανάγκες ε, που εντοπίζουν. Τώρα, το θέμα της αξιολόγησης επίσης είναι σημαντικό. Ο αξιολογητής δεν θα πρέπει ε, να δρά στον τομέα της αγοράς, αγορά προς αγορά, market to market, όπως είναι το usage, ε, σχεδόν πέρασε το πεντάλεπτο. Τι να σας πω, για τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Ξέρουμε ότι αυτά είναι άλλα ζωάκια, αλλά ε, υπάρχουν και ερωτήματα εκεί, πολύ σημαντικά που δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Η σύγκρουση συμφερόντων, ακόμα και στο στάδιο πριν γίνει εξαγορά. Ποιο ενημερώνεται για ποιο θέμα και ποιο έχει πρόσβαση σε τι. Και η υπερβολική μόχλευση ε, είναι επίσης ένα ζήτημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί και έχει σημασία. Και τέλο κάτι για τη ε, κυβέρνηση την εταιρική, corporate governance. Οι επενδυτές, εκτιβιστές επενδυτές, ε, έχουν αναλάβει κάποια δράση, αλλά δεν έχει δοθεί απάντηση. Δεν είναι μόνο εταιρικό δίκαιο εδώ το δίκαιο που ισχύει. Σκεφτείτε το σας παρακαλώ. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Να συμμετέχουν και οι μέτοχοι. Αυτή τη στιγμή η κυριαρχή αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η έκθεση Walker και πρέπει να γίνει δουλειά. Εκεί έχω ξεπεράσει το χρόνο μου κατά ένα λεπτό. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιη ότι κάποια από αυτά τα θέματα θα τα ξανασυζητήσουμε την ώρα των ερωτήσεων. Και συνεχίζουμε πάρα πολύ γρήγορα. Προχωρούμε στον επόμενο μιλητή μας που είναι ο κύριος Ρόμπιν ε, Όλιβερ. Α, περνούμε τώρα στις τρίτες χώρες και στους αιματοφύλακες. Έχουμε τον κύριο Ρόμπιν Όλιβερ, λοιπόν, που είναι επικεφαλής της EMA Compliance στην τράπεζα State Street. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, Ρόμπιν. Και Πάλι θα βάλουμε το χρονόμετρο. Uh, Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ευχαριστώ τα μέλη τη Επιτροπή για την ευκαιρία που μου δίνουν ε, να καταθέσω εξ ονόματο State Street, κυρίω για τι τρίτε χώρε. Ε, είμαι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση για την Αφρική και η έδρα μας είναι στη Βοστόνη και έχουμε ισχυρή πανευρωπαϊκή παρουσία σε 27 χώρες είμαστε και σε 100 αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο 13,33 δολάρια σε στοιχεία ενεργητικού παρακολουθούμε ε, και διαχειριζόμαστε 1,7 δισεκατομμύρια. Έχουμε συνεργάτες σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα μου ζητήθηκε να καλύψω τρία συγκεκριμένα τμήματα από την προοπτική των τριτών χωρών. Η, ευθύνη των θεματοφυλάκων, η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων. Ε, και τα επενδυτικά σχήματα οι διασυνοριακές επενδύσεις είναι, είμαστε υπέρ των διασυνοριακών επενδύσεων και οι εκθέσεις για συστημικούς κινδύνους σε διάφορες αγορές είναι κάτι πάρα πολύ λογικό. Τα σχόλια περί δέωσα επιμέλειας με βρίσκουν σύμφωνο τα σχόλια που ακούσαμε από πλευρά Caesar. Για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και τον προσδιορισμό των ευθυνών ακούστηκαν θετικά σχόλια και θέλουμε να υπάρχουν ανεξάρτητοι θεματοφύλακες. Ε, η γενικότερη καταχώρηση των διαχειριστών των εναλλακτικών επενδυτικών ταμείων είναι κάτι το ευκταίο κυρίως στις τρίτες χώρες. Υπάρχουν κάποια στοιχεία της οδηγίας ε, που κατά τη γνώμη μας δεν μπορούν να εφαρμοστούν ως έχουν ε, και ε, πάσχουν σε μεγάλο βαθμό. Οπότε εμείς προτείνουμε μια προσέγγιση ε, που συμπεριλαμβάνει τα προηγούμενα που υπάρχουν στην κείμενη νομοθεσία και την τρέχουσα πρακτική στις αγορές ε, το καθεστώς για ΣΕΚΑ έχει λειτουργήσει αισίως όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει ε, και ε, σίγουρα θα συνεχίσει έτσι η κατάσταση οπότε θέλουμε να χρησιμοποιηθεί όσο μοντέλο και για την επικείμενη νομοθεσία. Το πρώτο κομμάτι που θα με απασχολεί στην παρέμβασή μου είναι η ευθύνη των θεματοφυλάκων ε, και ε, ε, πρόκειται για μία από τις μονάδες που φροντίζουν τα στοιχεία του ενεργητικού των επενδυτών και η διαχείριση των ε, στοιχείων ενεργητικού που έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής από τέτοιες μονάδες custodian ε, ήταν καλή ε, και θεωρούμε ότι είναι δυσανάλογα μεγάλη αντίδραση για τους διαχειριστές των ελλακτικών επενδυτικών ταμείων μετά από τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν μιλώντας ε, για τους κινδύνους τώρα των ε, συμμετεχόντων που ε, φεύγουν από την αγορά και κίνδυνοι λόγω της συγκέντρωσης ή άλλοι συστημικοί κίνδυνοι θα οξυνθούν εάν ορίσουμε αυστηρά ποιος φέρει την ευθύνη κυρίως στον τομέα των συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι επενδυτές είναι σημαντικό ε, να έχουν στη διάθεσή τους τέτοιες ε, μονάδες καστόντιαν ε, όταν μιλάμε για άκρος κεφαλοποιημένες εταιρείες, επενδύσεις δηλαδή σε μεγάλη κλίμακα. Ε, θεωρούμε ότι μειώνεται η προστασία των επενδυτών και αυξάνεται το κόστος αν εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις ε, της οδηγίας ε, όταν χρειάζονται, όταν λειτουργούμε μάλλον όλοι σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Νομίζω ότι θα πληγούν οι ίδιοι οι επενδυτές. Τώρα θεωρούμε ότι για οποιονδήποτε διαχειριστεί το θέμα του θεματοφύλακα είναι ένα κόστος που πρέπει να καταβάλει. Οι δραστηριότητες ε, δέουσας επιμέλειας θα είναι χρήσιμες ε, για μας και τα πρότυπα σχετικά με την ε, επανόρθωση των ε, μη αιτιολογημένων ζημιών ε, υπακούν σε ένα σύστημα που έχει λειτουργήσει καλά μέχρι στιγμής και δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων τώρα, delegation, είναι σημαντικό για μας ε, σε επίπεδο θεματοφύλακη, σε επίπεδο αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού, σε όλη την αλυσίδα, σε παγκόσμιο επίπεδο να μπορούμε να εκχωρούμε αρμοδιότητες, γιατί έχουμε παίχτες σε διάφορες αγορές που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε το κόστος και να προσφέρουμε ε, ε, υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας. Θέλουμε να υπάρχει ενεργός εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δεν ε, κρίνουμε ότι πρέπει να περιορίζεται αυτό μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να περιοριζόμαστε σε μία μόνο εκχώρηση αρμοδιοτήτων. και ήδη παρέχουμε ε, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ε, για τη δέωσα επιμέλεια και θα συνεχιστούν αυτές οι δραστηριότητες μας ε, για οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού έχουμε υπό τον έλεγχό μας. Και θα θέλαμε διευκρίνη σχετικά με τα πρότυπα που πρέπει να εφαρμοστούν για τη δέωσα επιμέλεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός, γιατί προς το παρόν υπάρχει μια σάφια. Τελευταίο κομμάτι, οι ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι σημαντικό για μας να τονίσουμε ότι παρότι κατανοούμε και τον λόγο για τον οποίο ζητείται ευρωπαϊκό διαβατήριο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κλάδους που δεν απαιτείται στο παρελθόν. Θεωρούμε το καθεστώς των ιδιωτικών επενδύσεων κάθε κράτος πρέπει να συνεχίσει να ισχύει ως έχει, διότι θα πρέπει να, συνεχιστεί, να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως και στο παρελθόν και ξαναλέω και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει και για τους διαχειριστές των επενδυτικών κεφαλαίων και για τα ίδια τα επενδυτικά κεφάλαια. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν για τους επενδύτε να έχουν πρόσβαση στα επενδυτικά κεφάλαια όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο κόσμο. Βέβαια, αν ε, ε, υπάρχει επαγγελματική και σωστή διαχείριση, ο περιορισμός των επιλογών ε, λόγω της συγκυρίας θα πλήξει τους επενδυτές γιατί λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου η κερδοφορία είναι πάρα πολύ σημαντική και όπως σας είπα και προηγουμένως λειτουργούν αισίως οι ισχύουσες διατάξεις. Θα θέλαμε να συνεχιστούν λοιπόν τα καθεστώτα ιδιωτικών επενδύσεων όπως και στο παρελθόν. Τέλος, έχουμε μια ανοιχτή αγορά προς το παρόν που λειτουργεί καλά Ίσως χρειάζεται ρύθμιση σε κάποια τμήματα σε μεγαλύτερο βαθμό και θα υποστηρίξουμε αυτές τις ε, προσπάθειες αν γίνουν καθόλου και τυπικά εντάξει αλλά ε, πρέπει να παραμείνουν ανοιχτέ οι επιλογέ των επενδυτών για να μην ε, επισύρει αυτό, ε, για να ελαχιστοποιηθεί μάλλον το κόστο διαχείριση των ιδιωτικών επενδύσεων. Σα ευχαριστούμε. θα ήθελα. Να εξηγήσω ότι ο Ρόμπιν είχε 10 λεπτά στη διάθεσή του, όχι 5. Από ό,τι Ε, δεν εξήλυσε το χρόνο του. Στη συνέχεια θα δώσουμε περισσότερο χρόνο στις απαντήσεις. Ερχόμαστε στην επόμενη ενότητα που θα διερευνήσουμε και είναι η άποψη από την πλευρά των πωλήσεων αλλά και των αγορών. Και θα ακούσουμε τον Άντωνι Μπέρν, στον οποίο είχαν επίσης δοθεί 10 λεπτά, αλλά θέλει να μιλήσει λιγότερο. Και έτσι θα έχουμε περισσότερο χρόνο για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σας. Λοιπόν, Πέντε, έχει. πέντε. Ναι, γιατί έχουμε δύο μιλητέ. Ναι, ναι, εγώ κάνω λάθο, λέει η πρόεδρο. Ναι, εσεί έχετε πέντε λεπτά και πέντε λεπτά ο κύριο Μάρκο Μίντερχοφ. Δεν μπορώ να διαβάσω τα χαρτιά μου εδώ πέρα. <laughs> Ζητώ συγγνώμη. Πέντε λεπτά, Άντωνι Μπέρν. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λέγομαι Άντωνι Μπέρν και εργάζομαι στην Deutsche Bank. Θα σας μιλήσω σήμερα για την πλευρά των πωλήσεων. Έχω κάνει μια σύνοψη θα σας μιλήσω πέντε λεπτά σε τρεις ενότητες. Πρώτα, σύντομα θα σας εξηγήσω τι είναι το prime brokerage, η μεσητεία δηλαδή, μετά το IFMD ε, θετικά και ανισχυτικά και στη συνέχεια ε, θα αναφερθώ στον εισηγητή τον κύριο Γοζές ε, απαντώντας σε ερωτήσεις τους. Τι είναι το prime brokerage, είναι η μεσητεία και καλύπτει πολλούς τομείς, το clearing, τη θεματοφυλακή, τις υπηρεσίες ενεργητικού, ε, αναφορές για τους πελάτες, χρηματοδότηση, security και πολλά ακόμα. Διαχείριση κινδύνου και παροχή συμβουλών. Θα πρέπει να εξασφαλίζουμε μία απόδοση λογική ε, για να ε, μπορεί το ταμείο που είναι πελάτης να πληρώνει τα δάνειά του. Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, οι απώλειες πιστώσεων από το prime brokerage lending, τη μεσητεία ήταν πολύ χαμηλές και έτσι μπορούμε να πούμε ότι δούλεψε το σύστημα πολύ καλά. Ως επενδυτής, ε, ο μεσίτης αυτό που ενδιαφέρεται είναι να έχει έλεγχο του ενεργητικού και ε, να πληρώνονται τα δάνεια, να αποπληρώνονται τα δάνεια. Ε, καλή ρύθμιση του κλάδου είναι σημαντική, ε, για μειώνεται έτσι ο συστημικός κίνδυνος και ε, καλύπτεται καλά η αγορά. Θετικά και αρνητικά τώρα σε σχέση με την οδηγία. Ο κλάδος μας υποστηρίζει πλήρως τους γενικούς στόχους της οδηγίας για να υπάρχει εστίαση στο συστημικό κίνδυνο, στην προστασία των επενδυτών και την αναρμόνιση στην Ένωση. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα συνολικό συνεκτικό σύστημα ε, και αυτό το έχουν πει και η G20 και η ΑΙΟΣΚΟ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμείς είμαστε υπέρ της καταχώρησης των manager hedge funds, ε, το να γνωρίζουν οι ρυθμιστικές αρχές ε, στοιχεία για το συστημικό κίνδυνο, ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο και ενισχυμένη διαφάνεια. Ο στόχος λοιπόν ε, της παρουσίασης είναι να εστιάσουμε ε, στους τομείς που χωρούν ε, βελτίωση. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θα σας τα φέρω επιγραμματικά και τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε. Οι θεματοφύλακες, depositories, αναβάλουν κάθε ευθύνη για τον κίνδυνο και τις απώλειες που δεν μπορούν να ελέγξουν. Αυτό σημαίνει όμως μεγαλύτερο κόστος και απώλεια ε, ε, σε επενδύσεις σε πολλές αγορές εκτός της Ένωσης. Ε, σε μεγάλο βαθμό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους επενδυτές αυτό. Δεύτερο στοιχείο, το μάρκετινγκ και κριτήρια αντιστοίχησης. Μεταξύ άλλων, οι επαγγελματίες επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό των καλύτερων μάνατζερ στον κόσμο. Ε, οι περιορισμοί στη μόχλευση θα έχουν αρνητικό ε, αποτέλεσμα, θα περιορίσουν, θα έχουν συγκριτικό μειονέκτημα και θα περιοριστεί η ε, δυνατότητα δράση μας. Απαντώ τώρα σε ερωτήσεις του κυρίου Γκοζές. Τι είναι ο ορισμός του prime brokerage, της μεστίας είναι η βασική μέθοδος με την οποία ο κλάδος ε, ασχολείται με ε, τη θεματοφυλακή, με την αναφορά. Δυστυχώς όμως δεν αναγράφεται στα κείμενά σας. Υπάρχει μια σύγκρουση στη χρηματοδότηση με το θεματοφύλακα. Οι επενδυτές περιορίζουν τον κίνδυνο με ε, διαφοροποίηση, με ανάλυση του κινδύνου, και ε, τη χρήση πολλών ε, brokers και custodians. Δυστυχώς ε, στην οδηγία αυτό δεν επιτρέπεται. Στη συνέχεια είπατε τι συμφωνίες υπάρχουν με το AIFM, AIF και τους βασικούς μεσίτες που είναι οι θεματοφύλακες του AIF. Σε όρους ειδικού χρηματοδότησης Έχετε ένα παράρτημα στο σημερινό κείμενο που αναφέρει αναλυτικά ε, το περιεχόμενο, το στάνταρ περιεχόμενο και το αντικείμενο ε, της συμφωνίας. Εμείς έχουμε εποπτεία από την Buffen FSA και SSA ε, στη Deutsche Bank. Έχουμε εσωτερικό λογιστικό έλεγχο και εξωτερικό κάθε τρεις μήνες. Τέταρτη ερώτηση αφορά το πώς ενημερώνονται για τον κίνδυνο οι ρυθμιστές. Με χαρά να σας δώσουμε και άλλα στοιχεία, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο κατά πόσο είναι χρήσιμα τα στοιχεία ε, ενοποιημένα και η παρουσίαση για να μην ε, είναι αυτό εις βάρος των επενδυτών. Η ΆΙΜΑ και η HFSB πάντα ενθαρρύνουν ε, τη σωστή αποκάλυψη κινδύνου. Τώρα, ποιε ε, είναι άλλε νομικέ ε, υποχρεώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να ε, θεσπιστούν. Είναι πολύ μεγάλη η ρύθμιση έτσι και αλλιώ στον κλάδο και αν θέλετε να συζητήσουμε και για άλλα μέτρα δεν διαφωνούμε. σα. ευχαριστώ για την ευκαιρία που, είχατε, που μας δώσατε συγγνώμη να ακουστεί η φωνή της Deutsche Bank σε αυτό το κλάδο. Ευχαριστώ πολύ. Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση περνούμε στον επόμενο μιλητή που είναι ο Μάρκος Μίντερχοφ ε, Γενικό Σύμβουλο στην Ευρώπη από την ε, Alliance Global Invest Europe, εταιρεία περιορισμένη ευθύνη. Είμαι ο Μάρκος Μίτερχοφε. ασχολούμαι με τη συμμόρφωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Alliance Global. Ε, για την εταιρεία μου θα έλεγα ότι είμαστε από τους ε, λίγους πραγματικά παγκόσμιους διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού στην Ευρώπη, με έδρα στην Ευρώπη. Έχουμε ισχυρή παρουσία στη ΣΥΠΑ και σε όλες τις μεγάλες αγορές της Ευρώπης αλλά και της Ασίας και Ειρηνικού. Όταν, ε, δείτε, όταν είδαμε την οδηγία για τους διαχειριστές των εναλλακτικών ταμείων, δεν την εξετάσαμε από την οπτική γωνία των hedge funds, ε, γιατί δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ούτε στα προϊόντα που προσφέρουμε, ούτε ε, για τους επενδυτές μας παρουσιάζουν ενδιαφέρον, γιατί οι πελάτες μας είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες της, του ομίλου Allianz, που ε, επενδύουν σε τομείς όπου δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία τα hedge funds. Οπότε για μένα το βασικό ζήτημα ήταν η οδηγία και το βασικό ζήτημα της οδηγίας για του διαχειριστές ήταν ο ορισμός ούτω ώστε να καλύψουμε όλους τους φορείς πέραν των ΟΣΕΚΑ ε, που καλύπτει και πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου όλα τα μη ευρωπαϊκά συλλογικά επενδυτικά σχήματα. Αυτό μας οδηγεί σε πάρα πολλές δυσκολίες στον ομιλό μας, γιατί όπως σας είπα στην αρχή έχουμε οργανωθεί σε παγκόσμια βάση και προσπαθούμε να έχουμε την καλύτερη πραγματογνωμοσύνη από εμπειρογνώμονες κάθε κλάδου, ε, από εμπειρογνώμονες της επιχείρησης και να φέρουμε αυτή την τεχνογνωσία στην Ευρώπη και αυτό γίνεται δυσκολότερο και σε ενίοτε αδύνατο αν παραμείνει όσο έχει αυτή η οδηγία για τους διαχειριστές. Ε, θα σας δώσω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα ε, που έχει παραβλεφθεί εντελώς στη συζήτηση. Εκτός Ευρώπης, ε, τα επενδυτικά ταμεία που βρίσκονται στην Ασία ή στον Ειρηνικό, που δεν είναι ως ΕΚΑ και θα υπάγονται στην οδηγία για τους διαχειριστές. Ωραία ως προς τη ρύθμιση τους θα υπακούν ε, στους κανόνες της, ε, τους εθνικούς, της εθνικής νομοθεσίας. Ε, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμένα ναι, τα γραφεία μας από τη ΣΥΠΑ, αλλά... Έχουμε και τους πελάτες μας στην Ασία και στον Ειρηνικό και θα, θα έχουμε ακολουθήσει τη λανθασμένη προσέγγιση. Και το ίδιο ισχύει για τις επενδύσεις των Ευρωπαϊκών Ταμείων, γιατί εκεί χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία εμπειρογνωμόνων που βρίσκονται σε άλλα μέρη του κόσμου για να σχολιάσουμε την ποιότητα των προϊόντων και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρουμε. Δηλαδή θα πληγούν τα αποτελέσματα για τους πελάτες μας. Ο Όμιλος Αλιάνς που είναι ο βασικός μας πελάτης θεωρεί ότι τελικά τελικά η προστιθέμενη αξία είναι ε, η αυτή η τεχνολογία που χρειάζεται για τον ασφαλιστικό τομέα και κυρίως για τις ασφάλειες ζωής. Όπως ακούσαμε και στην προηγούμενη συζήτηση, ένα καθεστώς για τις ιδιωτικές επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτο γιατί είναι ένα εργαλείο που θα προσδώσει νομική ασφάλεια σε ένα σύστημα ε, ε, εξαιρετικά κατακαιρματισμένο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αν αυτό είναι ο στόχος ε, για τον οποίο προτείνεται αυτό το σύστημα, αυτό το καθεστώς των ιδιωτικών επενδύσεων, θα το υποστηρίξουμε. Και θα υποστηρίξω και αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου εδώ δίπλα, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτό να είναι ένα κίνητρο για να καταργηθούν τα εθνικά επενδυτικά σχήματα, τα οποία λειτουργούν μια χαρά και δεν χρειάζεται να περιορίσουμε τις επιλογές των επενδυτών. Τελευταίο σημείο. Το θέμα των θεματοφυλάκων που αναφέρθηκε από τους συναδέλφους μου, από την πλευρά της αγοράς ε, της εξαγοράς τίτλων. Θέλουμε οι τιμές ε, για τις υπηρεσίες ε, ε, φυλακής, custodian services, να παραμείνουν σε λογικό επίπεδο και όπως ακούσαμε υπάρχει μία επίπτωση σε παγκόσμιο επίπεδο και ελοχεύει ο κίνδυνος κάποιες αγορές να μην είναι διαθέσιμες πλέον ως επενδυτικές αγορές αν εφαρμοστεί αυτό το αυστηρό καθεστώς προσδιορισμού της ευθύνης και όπως είπε και ο Ντιβάιμερς, ε, τελικά δεν μπορεί κανεί να επιχειρηματολογεί και να λέει ότι το καθεστώς των ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να είναι λιγότερο αυστηρό σε σχέση με το καθεστώ για τους διαχειριστές γιατί θα έχουμε spillover, προφανέστατα. Και πρέπει να γίνει θεμελιώδης ανάλυση των δεδομένων και θα κλείσω με αυτή την παρατήρηση δεν θεωρώ ότι αυτό το θέμα είναι θέμα μόνο επενδυτικών ναι, κεφαλαίων. Πρόκειται για παγκόσμιο καθεστώς ε, φυλακής, καστόντιαν ε, ε, φύλαξης. Ευχαριστώ. Thank you very Σας ευχαριστώ πολύ. Μάρκος. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενη ενότητά μας που είναι πάλι δύο μιλητές για τα συνταξιωτικά ταμεία pension funds. Πρώτη ομιλή Πρώτος ομιλητής είναι ο Κρίς Ντούμα, επικεφαλής ε, της υποστήριξης επενδύσεων και Active Ownership. Πού είστε, α, και έχετε το λόγο. Well, thank you uh, uh, for the invitation to, to speak at this uh, hearing. MN Services is a... Καλημέρα σας. Ε, ε, εγώ ασχολούμαι με τη διαχείριση του ενεργητικού οικοσυκλάδων. Ε, περίπου ε, και αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινούμε και πάνω σε αυτό μιλάω. Θα ήθελα να, απευθυνθώ, να σας απευθύνω τέσσερα θέματα. Το ένα είναι ε, η γενική διαχείριση, το δεύτερο είναι η ευθύνη των θεματοφυλάκων, το τρίτο είναι τι προκαλεί τους κινδύνους, οι οργανώσεις ή η συμπεριφορά και το τέταρτο αφορά το ε, φορτίο που θα πέσει στα συνανταξιοδοτικά ταμεία σε σχέση με, ορισμένους, με ορισμένες εναλλακτικέ επενδύσεις. Καταρχήν λοιπόν, ο στόχος της οδηγίας ποιο είναι, ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν απολύτως δίκιο που απευθύνουν αυτό το θέμα το οποίο βασίζεται στα διάφορα επενδυτικά ταμεία στην απαρχή του και συμφωνούμε με την αρχή γενικά αυτής της οδηγίας αλλά πρέπει να πούμε ότι ένας από τους στόχους είναι η προστασία των επενδυτών και όπως ξέρετε όλοι εδώ ότι υπάρχει ένας τρόπος ε, να ακολουθούνται διάφορες διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου και σε πολλές περιπτώσεις σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη αυστηρότητα στην πράξη από ό,τι προτείνεται τώρα στην οδηγία. Η οδηγία βεβαίως μπορεί να βοηθάει σε ορισμένες απόψεις αλλά πρέπει να είναι σαφές ότι οι επαγγελματίες επενδυτές εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα και ελέγχους και διαδικασίες πιο αυστηρές από ό,τι προτείνεται στην οδηγία. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το να εξετάσουμε ε, τι ε, ε, προκαλεί αυτό το συστημικό κίνδυνο και έτσι ε, πρέπει να εστιαστούμε στο περιεχόμενο και στην ε, συμπεριφορά ορισμένων βιομηχανιών ειδικά για τις εναλλακτικές επενδύσεις οι οποίες αφορούν όλες τις πλευρές της χρηματοοικονομικής αγοράς και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, δεν τονίζεται ιδιαίτερα στην οδηγία. Θέλω να σας δώσω μερικά μικρά παραδείγματα. Το ένα είναι ότι θεωρούμε καταρχήν το θέμα του empty voting σαν ε, περίπτωση κινδύνου συστημικού. Γίνεται μια σαφής διάκριση του οικονομικού κινδύνου και επίσης αυτό που είναι, έχει τα δικαιώματα στις ε, μετοχές ε, σε σχέση με το επενδυτικό ταμείο. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν συστημικό κίνδυνο οπωσδήποτε. Βλέπουμε ότι σωστά η αμοιβή είναι ένας στόχος ε, που απασχολεί πολύ τις τράπεζες και ε, πολλές φορές το θέμα της αμοιβή στην ε, βιομηχανία τη σχετική μπορεί να δημιουργήσει συστημικούς κινδύνους και πρέπει να ασχοληθεί ο τραπεζικός τομέας μαζί του όπως και εμείς. Το τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι ότι υπάρχουν φήμες ότι η Σουηδική Προεδρία ε, θα κάνει ορισμένες ε, μοχλεύσεις ε, και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ κακό παράδειγμα και προηγουμένο γιατί είναι μια περίπτωση όπου χρειαζόμαστε μια συνολική βάση για τη μόχλευση και όχι μόνο να δούμε τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν θα ήθελα να βγει από την οδηγία γιατί εδώ η οδηγία μας βοηθάει και άλλες ε, ορισμένες παρατηρήσεις στο θέμα του φορτίου. Πρέπει να εξηγήσω ότι πρέπει να έχουμε πολλές φορές αντιμετώπιση πολύ μεγάλων πελατών οι οποίοι κάνουν τις δικές τους ε, επενδύσεις και έχουμε μικρά, ε, μικρότερα συνταξιωτικά ταμεία και για αυτά τα μικρότερα ταμεία είναι ειδικέ αγορές, στοχευμένες αγορές όπου πρέπει να δούμε πώς θα μπουν στη χρηματοοικονομική αγορά για να έχουν μια θέση εκεί πέρα την οποία δεν έχουν ε, τα μικρά συνταξιοδοτικό ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω χήματα θα ε, μπουν στο εύρος των ε, συνταξιοδοτικών ταμείων. Νομίζω ότι υπάρχει μια εξαίρεση η οποία παρέχεται για τις συντάξεις και για το μέσο που χρησιμοποιείται για τα συνταξιοδοτικά ταμεία που τους δίνεται έτσι το δικαίωμα να πάρουν μέρος στη χρηματοοικονομική οικονομική αγορά. Και η τελευταία παρατήρησή μου σε αυτόν τον τομέα είναι ότι η οδηγία όπως έχει τώρα ε, προτείνει μια, ένα περιορισμό, πολύ σοβαρό περιορισμό των συνταξιδοτικών ταμείων στην επένδυση των ευρωπαϊκών ταμείων και επενδύσεις που κάνουμε για τους πελάτες και για τις υπηρεσίες μας είναι εκτός των ταμείων της ΕΕ και μας ζητούν ε, καταγραφή μέσα στην ΕΕ και αναγνώριση. Αυτοί δεν είναι βέβαια οι ίδιοι οι οποίοι έχουν τα υψηλά προσόντα, τα ταμεία εκείνα τα οποία είναι, ε, ε, έχουν πολύ καλή αξιολόγηση μέσα στον όμιλο. Έχουν περιορισμένες λοιπόν δυνατότητες αυτά τα ταμεία και δεν μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις στα ευρωπαϊκά ταμεία κάτι το οποίο θα ήταν ενδεχομένως αντίθετο προς τα συμφέροντα όσων επενδύουν στον τομέα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο συνταξιδιωτικό ταμείο για το της συμμόρφωσης Ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημερινή ακρόαση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ενώπιόν σας. Ε, θα συμφωνήσω με του προλαλήσαντες σε μεγάλο βαθμό ε, και άρα μπορώ να είμαι και πολύ πιο σύντομος. Ε, καλό και για σας. βέβαια θα είμαι λίγο πιο αρνητικός και αυτό συμπίπτει και με την αξιολόγηση αντικτύπου και τα συμπεράσματά της που είδαμε χτες για αυτή την οδηγία συγκεκριμένα. Για να μην υπάρχει επικάλυψη και επειδή δεν έχουμε έχουμε χρόνο θα περιορίσω την, την παρουσίαση μου ε, στον, ε, σε μια έκκληση ουσιαστικά να, όλα τα θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο να ακολουθήσουν ε, την προσέγγιση τη καλύτερη νομοθεσία. Όλοι επιθυμούν νομοθετική ρύθμιση, αλλά οι αρχέ καλύτερη νομοθεσία δεν πρέπει να παραβλεφθούν γιατί αυτή η οδηγία μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ την ευμερία των επενδυτικών ταμείων. 1,4 δις σε κόστος συμμόρφωσης να ε, ή επίσης αύξηση ε, των ε, ασφαλιστικών εισφορών λόγω της σπεσμένης αυτής νομοθεσίας. Δεν είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Ε, εν είδη ιστορικού υποβάθρου να σας πω ότι διαχειριζόμαστε επενδυτικά ταμεία και έχουμε 1,33 ε, το χρόνο σε διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και ε, εκπροσωπούμε και εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία. Λειτουργούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, 57% παρουσία στη ΣΥΠΑ και το υπόλοιπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αναδυόμενες αγορές μόνο 8%. Συνολικά ε, ε, έχουμε 70 με 80% στοιχείων ενεργητικού που οι ίδιοι διαχειριζόμαστε το δικό μας χαρτοφυλάκιο και τα προϊόντα και οι περιοχές που χρειάζονται συγκεκριμένη τεχνογνωσία ανατίθενται εξωτερικά σε ε, διαχειριστές. Οπότε αν εισαχθούν αυτοί οι περιορισμοί θα έχουμε πρόβλημα με την επιλογή των διαχειριστών και θα έχουμε πρόβλημα με το χαρτοφυλάκιό μας και το ίδιο και οι θεσμικοί επενδυτές κυρίως σε αναδυόμενες αγορές σε νέα προϊόντα και ε, στην τήρηση των ε, νομοθεσιών περιβαλλοντικών ε, και άλλων. Η πρόταση που τώρα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο είναι μια καλή πρωτοβουλία, το αναγνωρίζουμε, αλλά αυτό όλα στην τωρινή μορφή τη. έχει περισσότερα αρνητικά παρά θετικά. Και... Αυτό είναι μοναδικό στην ευρωπαϊκή ιστορία διαχείρισης και ελέγχου των αγορών. Και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν συμφωνήσει ομόφωνα στα 42 μέτρα. Γιατί η Ευρώπη λοιπόν είναι τόσο καινοτόμα στο ΜΕΦΙΤ, στο γιουσίτς και τόσο ε, ομόφωνη. Κατά την άποψή μου, είναι ότι ε, πραγματικά αυτό που ευνοείται από τις μίσεις αυτές είναι ο κλάδος. Και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η οδηγία αλλάζει δρόμο και επιλέγει τον οδό της διαφάνειας. Εμείς ε, θεωρούμε ότι χρειάζεται ε, ανάλογη προσέγγιση, όχι απουσία διαβούλευσης, όχι τέτοιες πρωτοβουλίες όπως έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ολέθριε οι συνέπειε και τα συμπεράσματα όταν είναι ε, σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου ε, επιπόλαια, αποσπασματική και ε, προθύστερη και χωρίς διαβούλευση. Για το G20 θα πρέπει να είναι τα συμπεράσματα τα ίδια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Γι' αυτό υπάρχουν και συστάσεις. Δεν μπορεί ένα συμβαλόμενο μέρος να αποσυρθεί μονομερός από τις υποχρεώσεις του. Και δυστυχώς αν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο μειονέκτημα, να προχωρήσουμε σε συνεννόηση και σε διάλογο με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Τελικά ε, θα επιβαρύνει με κόστος, με χαμηλή απόδοση τα χαρτοφυλάκια και πολύ Ευρωπαίοι, εκατομμύρια Ευρωπαίων θα πληγούν ε, που συμμετέχουν σε συνταξιδοτικά ταμεία. Με τη γύραση του πληθυσμού και τη συρρήκνωση της οικονομίας, τη μεγάλη ανεργία, ε, την κρίση, ε, τον πληθωρισμό, το χρέος. Δεν μπορούμε να αποτύχουμε στην οδηγία αυτή. Δεν έχουμε περιθώρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ρωτώ, τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσιλωμένα σε αυτή την οδηγία. Θέλουν να ακολουθήσουν την αρχή τη καλύτερη ρύθμιση για τα προϊόντα και τα παράγωγα, γιατί με τις ε, προτάσεις τους δεν εξυπηρετούν την αγορά. Για την ε, διαφάνεια και τις διαβουλεύσεις δεν μας έχετε ρωτήσει ποτέ μας τους επενδυτές. Γιατί τα κάνουν αυτά ε, ε, στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου με μεγάλη επιρροή καλά οργανωμένων λόμπι και αγνοώντας τις συστάσεις και του G20. Ως κλάδος λοιπόν θεωρούμε ότι θα πρέπει ε, να προχωρεί η διαφάνεια. Εμείς ό,τι έχουμε μάθει το έχουμε μάθει από διαρροή εμπιστευτικών και απορρίτων εγγράφων ε, τα τελευταία χρόνια. Πώς είναι δυνατό αυτά να ε, συνάδουν με την ακαιρεότητα που τώρα πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε διαπραγματευτής προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντα της ιδιαίτερης περιφέρειας. Αν θέλει κανείς να ξεκινήσει σωστά αυτή η οδηγία, γιατί να δεχόμαστε συμβιβασμούς χολούς και περίεργους ε, και ε, υπάρχει τέτοια διαφάνεια στην τόσο σημαντική ρύθμιση. Θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό το κοινοβούλιο, δεν μπορεί να προέρχεται από το σκότος μια οδηγία και να επικαλείται τη διαφάνεια στη χάραξη πολιτικής. Θα πρέπει και η ποιότητα της οδηγίας αυτή να βελτιωθεί και θα βελτιωνόταν εάν ε, το Κοινοβούλιο καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει προσωρινά αυτή την οδηγία γιατί θα έρθουν πολλές τροπολογίες και μέχρι το καλοκαίρι να φέρει καλύτερη πρόταση με ευρύτατη διαβούλευση και ε, τους επενδυτές, τα συνδοξιωτικά ταμεία και αυτούς που είναι άμεσα πληγόμενοι και ενδιαφερόμενοι και δεν έχουν ε, συμμετάσχει. Καλώς. Σταματώ εδώ. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα διαβάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε τώρα να δείτε ότι θα υπάρξει πίεση για να συνεχίσουμε ε, και Επίσης έχω ένα κόκκινο φωτάκι το οποίο μου λέει ότι οι διερμηνείς βρίσκουν ότι μιλάτε λίγο γρήγορα, έχουν, ε, δεν έχουν το κείμενα μπροστά τους. Ας περάσουμε τώρα ε, στα συνδικάτα και έχουμε τον πρώτο μιλητή την Τζάνετ Βίλιαμσον, η, η οποία πήρε μέρος στο Trader Unions Congress. Ε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου βάλετε σήμερα ε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την συνάδελφό μου. Θα ήθελα να αρχίσω από το κλειδί του UC, ε, από τους στόχους. τη καταρχήν ο κανονισμός θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος και πολύ αυστηρός σε σχέση με τον χρηματοοικονομικό τομέα συνολικά. Θα πρέπει να προστασεύει τους εργαζόμενους και τα συμφέροντά τους σε εταιρείε οι οποίες επενδύουν ή αγοράζουν στο FMI. E. Ε, επίσης θα πρέπει να υπάρχει ε, μια, ισο, μια ισοτιμία ε, και πιστεύουμε ότι ο χρηματοοικονομικός τομέας εξυπηρετεί τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, δεν συμβαίνει το αντίθετο και αναγνωρίζουμε ότι το θέμα της ισοτιμίας είναι κάτι που έχει σχέση με την βασική αρχή ε, που πρέπει να διέπει την, ε, ε, τον χρηματοοικονομικό τομέα συνολικά που έχει ορισμένους, ορισμένες αδυναμίες, ορισμένους επιμέρους τομείς. Θα πρέπει να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση και να εστιαστούμε στις, στις περιοχές κλειδιά. Θα ήθελα να πω τώρα δύο λόγια για το, την επίπτωση που έχει στους εργαζόμενους το θέμα της ισοτιμίας. Καταρχήν ένα θέμα κλειδί είναι ότι όταν υπάρχουν ε, διάφορα προβλήματα μετά από το γεγονός παρεμβαίνουμε συνήθως δεν γίνονται ορισμένες συζητήσεις ε, πρώτερες και πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει πρέπει να γίνει μια έρευνα και να γίνονται αναφορές ε, κάτι το οποίο υπάρχει σαν πλαίσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και το οποίο απασχολεί τα συνδικάτα στις μεγάλες εταιρείες Επίσης πιστεύουμε ότι υπάρχουν επικαλύψεις της και για, ε, πολύ συχνά και αυτές είναι μία αιτία της διαστρέβλωσης της ισοτιμίας. Υπάρχουν πολλές φορές ε, πανεπιστημιακές εργασίες σε αυτόν τον τομέα ε, και οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει πολλές φορές να πληρώνουμε και ειδικού που ανήκουν σε πανεπιστήμια για να μας δίνουν συμβουλές πάνω σε αυτά τα θέματα. Καταρχήν για το θέμα της προστασίας των συμφερόντων των εργαζομένων μπορούμε να πούμε ότι χαιρετίζουμε τα άρθρα 28 και 29 της οδηγίας ε, για το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου το οποίο μιλάει για ένα φορτίο το οποίο υπάρχει ε, σε αυτόν τον τομέα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα των καταστάσεων όπου χρειάζεται μια διαβούλευση σε τομείς κλειδιά για να μην χάσει από αυτό η εταιρεία για να δούμε επίσης το θέμα το οποίο είχα αρχίσει να σας αναπτύσσω πιστεύουμε ότι χρειάζονται ορισμένες προβλέψεις σε σχέση με την οδηγία οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται και στον τομέα της ισοτιμίας και οι συλλογικές συμφωνίες και οι σχέσεις μεταξύ των συνδικάτων θα πρέπει να γίνονται ε, σεβαστές. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο το οποίο ανάφερε και ο συνάδελφός μου να πω δύο λόγια καταρχήν για την αμοιβή και για τη θέση των συνταξιδοτικών ταμείων. Ε, τα TUC αποτελούν ένα δίκτυο χιλίων περίπου συνταξιδοτικών ε, ταμείων και επενδυτών οι οποίες ε, ζητούν ε, την προστασία των συμφερόντων τους και είδαμε ότι υπάρχουν αυτά τα συνταξιδοτικά ταμεία τα οποία μπορούν να επωφεληθούν από τις ε, ε, μελέτες οι οποίες ε, έχουν εκφραστεί σε ορισμένα άρθρα αυτής της οδηγίας. Επίσης πρέπει να τονίσουμε το ότι υπάρχουν ορισμένες διεκδικήσει σε σχέση με την ε, μείωση των αποτελεσμάτων των συνταξιοδοτικών ταμείων και γι' αυτό ε, θα πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτό της ε, και να αυξήσουμε το επίπεδο της προστασίας ούτως ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες επιστροφές από τις επενδύσεις των κεφαλαίων. Εάν ε, δείτε τι επιστροφές υπάρχουν σήμερα από το 1985 μέχρι το 2008 υπάρχουν ορισμένα ε, ταμεία τα οποία εξαγοράστηκαν και τα οποία βασίζονται σε ισοτιμίες που όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Οι, οι εναλλακτικές ε, επενδύσεις πιστεύουμε ότι τελικά έχουν μια αρνητική σχέση με την αύξηση και θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ε, προς αυτή την κατεύθυνση θα σταθώ εδώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ και εγώ και ο τελευταίος ομιλητής μας από τα συνδικάτα, από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων είναι ο Ρεν Χόφμαν. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο συνάδελφός... Η κυρία Τζάνετ Βίλιαμσον τα είπε πολύ ωραία και έδειξε ποιο είναι το ενδιαφέρον των συνδικάτων και του συνδικαλιστικού κινήματος για αυτή την νομοθεσία συγκεκριμένα. Εγώ προσωπικά θέλω να κάνω μερικά συμπληρωματικά σχόλια μόνο. Καλωσορίζουμε βεβαίως την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε επίγνωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχε αρνηθεί να κάνει πρόταση για ε, αυτά τα επενδυτικά ταμεία και συμφωνούμε με αυτό που είπαν και άλλοι ομιλητέ, ότι χρειάζεται καλύτερη ρύθμιση, καλύτερη νομοθεσία. Και όταν πρόκειται για αυτό το καλύτερο, είναι τεράστιε διαφορέ από εκεί και πέρα τι εννοεί ο καθένα όταν μιλάει για καλύτερη νομοθεσία και καλύτερε ρυθμίσει. Και ένα θέμα για το ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα είναι αρκεί αυτή η πρόταση να περιορίζεται στους διαχειριστές των ταμείων, των managers ή και τα ταμεία ολόκληρα, τα συνταξιοδοτικά. Θα πρέπει επίσης να αποφευθούν παραθυράκια στην νομοθεσία για να δώσουμε ε, ένα καλό παράδειγμα του ευνομοθετή. Χρειαζόνται τα κατόφλια που προτείνει η οδηγία ή το σχέδιο οδηγίας. 100 εκατομμύρια για τα hedge funds είναι αυτό το καιρό και 500 εκατομμύρια για τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Είναι απαραίτητα αυτά τα κατόφλια. Και... Ε, θα πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα παραθυράκια που σας είπα για τις εξαιρέσεις. Καλωσορίζουμε αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο οδηγίας για την πόλεις χωρίς αντίκρισμα θα πρέπει όμως να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη στην εξήγησή της ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέματα ρευστότητας και κεφαλαϊκές ε, ε, απαιτήσει, συγγνώμη, θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη. Η Τζάνετ αναφέρθηκε σε αυτά τα θέματα και στον αντίκτυπο που έχουν εναλλακτικά επιθετικά ταμεία στην απασχόληση και δεν μπορώ παρά να παραθέσω μια μελέτη που δεν έχουν κάνει τα συνδικάτα αλλά η Standard Poor's παρακαλώ που λέει ότι πάνω από η μισή ε, δραστηριότητα φέτος αφορούσε ε, τέτοια χαρτοφυλάκια και εταιρείε διαχείριση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τώρα, τι γίνεται με την ανεξάρτητη αξιολόγηση, με την καλύτερη διαχείριση των θεματοφυλάκων, ε, καλύτερη διαχείριση κινδύνου, καλύτερη ανάθεση, delegation και όλα αυτά που αναφέρθηκαν από άλλους ομιλητές. έλεγχος της μόχλευσης για να μην μειώνονται τα στοιχεία του ενεργητικού. Αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο για να βελτιωθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά θα συνεισφέρει και στην πραγματική οικονομία και θα περιορίσει ε, το εξωτερικό κοινωνικό κόστος και θα πρέπει να πάρουμε σαφή ε, παραδείγματα και διδάγματα από την κρίση, να μην επιτραπεί να υπάρξει ξανά τέτοια κρίση. Γενικά είμαστε προσυλλοβαίνει στο πλαίσιο του G20 και της συμφωνίας. Χρειάζεται βεβαίως καλύτερη νομοθεσία, καλύτερη ρύθμιση και το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρήθη ε, προβλημάτων, σφαλμάτων και θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση, να κάνει κάποιες προτάσεις που θεωρούμε ότι είναι κρίσιμες και να μείνει στα δικά του ψηφίσματα. Και πέρα από κομματικές ε, διαφορές. Συμφωνούν όλε οι πολιτικέ ομάδε σε αυτό. Αν θέλετε να κάνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις, με χαρά να σα τι δώσουμε. Thank you very much. Uh, we now have just... Ευχαριστούμε. Έχουμε λιγότερο από μία ώρα τώρα για τις ερωταπαντήσεις. Ζητώ από τα μέλη, διότι ως συνήθως έχουμε ένα μακρύτατο κατάλογο ομιλητών. Θα ζητήσω από τα μέλη λοιπόν να περιοριστείτε σε ερωτήσεις. Να μην προσφωνείτε ομιλίες παρακαλώ. Ένα λεπτό θα έχετε Καστός, και ε, θα δώσω λίγο περισσότερο χρόνο στον εισηγητή και σας προτείνω να ακούσουμε τον εισηγητή και τους σκιώδεις ή τους αναπληρωτές τους πρώτα και μετά τα υπόλοιπα μέλη που ζήτησαν το λόγο. Ζαν Πολ, ε, θα είχες ερωτήσεις προς εμπειρογνώμονες? Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα υποβάλω ερωτήματα, όχι γιατί δεν έχω, αλλά γιατί προτιμώ να αφήσω το χρόνο στους ε, συναδέλφους μου που θέλουν να εμβαθύνουν σε αυτό το ζήτημα. Μία παρατήρηση θα κάνω. Αρχίζοντας ε, τη συζήτηση είπα ότι καλή είναι η οδηγία, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως ακούσαμε. Πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Είμαστε σε διαδικασία συναπόφασης. Δηλαδή, πρότεινε ένα κείμενο η Επιτροπή και το Συμβούλιο τώρα και το Κοινοβούλιο πρέπει να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους σε ισότιμη βάση, απολύτω ισότιμη βάση με το Συμβούλιο. Αν δεν συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο δεν θα υπάρξει οδηγία. Σας διαβεβαιώ θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εγκριθεί η οδηγία. Αλλά στις σημερινές παρεμβάσεις ε, διευκρίνησαν όλοι κάποια ζητήματα και ε, τόνισαν κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες που υπάρχουν και ενίοτε έκαναν και προτάσεις ρύθμιση των προβλημάτων. Στις 25 Νοεμβρίου θα εκδώσω την έκθεσή μου αν όλα πάνε καλά και έχουμε και δύο μήνες για τις τροπολογίες μετά στη συζήτηση, της διαπραγματεύσης και για να προετοιμάσουμε τις συμβαστικές λύσεις που τον Απρίλιο θα υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει ολοκληρωθεί η δική μας εργασία και ε, ο Ισκιώδης και ο υποφαινόμενος δεν θεωρούμε ότι είναι άριστη η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, βέβαια, δεν είχαν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους. Ο αρμόδιος επίτροπο αντιστάθηκε σε μεγάλο βαθμό στο αίτημα του Κοινοβουλίου που ζήταγε ρύθμιση στην αγορά και για όλου αυτού τους λόγους επιδέχεται βελτιώσεις ε, η πρόταση της Επίτροπή και νομίζω ότι είναι κοινή μέρημνα όλων να έχουμε συγκεκριμένη και αποτελεσματική νομοθεσία που δεν θα παραλύσει τον κλάδο αλλά θα ελέγξει με αποτελεσματικό τρόπο του κινδύνου ε, που υπάρχουν και δεν μπορούμε να επικαλεστούμε μόνο την κερδοφορία, ε, γιατί είδαμε με την κρίση ότι κατέρευσαν διάφορα ιδρύματα και έθεσαν σε κίνδυνο ολόκληρη την οικονομία. Είναι συλλογική εργασία. Κύριε Γόφμαν, σα διαβεβαιώ, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια συμβαστική λύση για να περάσει αυτή η νομοθεσία, διότι είναι απαραίτητη. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή που θα μας εξετάσει το ρόλο του Κοινοβουλίου στο θέμα της ε, διαφάνειας σε σχέση με διάφορα άλλα θεσμικά όργανα. Κύριε Γκέμπελς, ο κύριος Γκέμπελς, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όπως και ο συνάδελφός μου θα ήθελα και εγώ να μη θέσω ένα ερώτημα αλλά να υποβάλω μερικά σχόλια σύντομα. Καταρχήν δεν ικανοποιήθηκα από αυτά που άκουσα γιατί οι περισσότερες παρεμβάσεις που είχαμε ήταν κάπως ε, δίπλα στο πλάι στον προβληματισμό δεν κάλυπταν τον προβληματισμό κατά την άποψή μου και μας λέγεται ότι ε, είμαστε υπέρ των μεγάλων αρχών στην αρχή όταν όμως ε, θα δούμε τα στα αυτό των μεγάλων αρχών μας λένε μην φύγετε τίποτα, μην αγγίζετε τίποτα ε, είμαστε εμείς οι επενδυτές οι επαγγελματίες και ε, κάνουμε τις επιλογές μας με μεγάλη φροντίδα κτλ. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση το ότι η κυρία Ρος μας είπε ότι δεν πρέπει να περιορίσουμε την ε, την ε, περίπτωση αυτή που μας απασχολεί ο κύριος Φρυς μας λέει ότι πρέπει να επιλέξουμε με μεγάλη φροντίδα τα ε, όρια αυτής της υπόθεσης και μας λέει ότι υπάρχει μια καθολική, μια παγκόσμια διάσταση σε αυτό το θέμα, ένα επίπεδο συνεκτικής ε, ε, επιθεώρησης, ενός συνεκτικού ελέγχου, ο οποίος δεν πρέπει να ασκεί διακρίσεις καθόλου. Βεβαίως, πολύ καλά. Λοιπόν, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, τελειώνω διαπιστώνοντας ότι ορισμένα από αυτά τα μεγάλα γεγονότα σημειώνονται ανάλογα με τις μεγάλες ρυθμίσεις. Αυτές οι επιπρόσθετες ρυθμίσεις είναι κατά των συμφερόντων των επενδυτών και των καταναλωτών. Θα ήθελα να σας πω ότι κυρία Πρόεδρε, πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι μου λένε γιατί τόσοι επενδυτές και τόσοι καταναλωτές έχασαν χρήματα γιατί τόσα συνταξιδιωτικά ταμεία βρίσκονται στο κόκκινο παρόλο που έχουν καταπληκτικούς επαγγελματίες και ειδικά στις κάτω χώρες, στις σκανδιναβικές χώρες, στη Μεγάλη ε, Βρετανία υπάρχουν τέτοια προβλήματα για τα συνταξιδιωτικά ταμεία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν επόμενο ο μιλητή θα επανέλθει, έχει βγει έξω. Παρακαλώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να περιορίσω τις ε, παρατηρήσεις μου σε δύο-τρεις σύντομες ερωτήσεις. Ε, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι για τις καταχρήσεις της αγοράς είδαμε μια διαφάνεια ε, και θα ήθελα να δω τι στοιχεία υπάρχουν για αυτήν την ε, δραστηριότητα σε σχέση με τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου. ποια είναι τα υπόλοιπα στοιχεία. Το δεύτερο ερώτημα έχει σχέση με την Deutsche Bank και την State Street όταν μιλάμε για τους κινδύνους των εγχειρημάτων προβλημάτων. Τι εάν ε, θέλουμε να ε, δούμε τις επιπτώσεις και προσπαθούμε να τις δούμε εργαζόμενοι ε, ποια είναι αυτά τα θεσμικά όργανα τα οποία απομένουν σε σχέση με τους θεματοφύλακες σύμφωνα με τη δική σας αξιολόγηση την ευθύνη των θεματοφυλάκων πόσο μεγάλα είναι αυτά και πόσο έχουν την δυνατότητα να πάρουν απεριόριστη ευθύνη θεματοφυλάκων είναι κοντά στα έξι και τι συστημικός κίνδυνο γνωστή τι συστημικοί κίνδυνοι προκύπτουν λόγω αυτού. Επίσης, ε, ποιο είναι το εύρος αυτών των δραστηριοτήτων. Ε, καταρχήν ε, υπάρχουν οι επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα μας απασχολεί σε σχέση με θέματα ανάπτυξης και το πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε περισσότερη ανάπτυξη σε περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο. σε ποια χώρα θα υπάρχει αποτελεσματικότητα αυτής της κλίμακας. θα ήθελα να έχω μια πιο καθαρή εικόνα. Και μια άλλη σύντομη ερώτηση σε σχέση με τις υπηρεσίες. Έχουμε ε, επίσης ε, ένα θέμα ανάληψης ε, του κινδύνου μόχλευσης. Ποιος θα αναλάβει τη μόχλευση σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα να ξέρω τι περιθώριο μας απομένει στην περίπτωση αυτή. Εάν έχουμε μία μόχλευση του κεφαλαίου στο στην ΕΕ, τι θα γίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ήθελα κάποια απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα πω στους εμπειρογνώμονες μου ότι αυτά τα θέματα πρέπει να τα έχετε σημειώσει σε ένα χαρτάκι, να τα έχετε στο μυαλό σας και να τα δώσετε στους σκιώδεις εισηγητές ε, πριν από την ε, αναχώρηση. Ο κύριος Σολεσμίτ, ναι, ο Δόκτωρ Φυσικά Κανείς εδώ δεν ζητά περισσότερη ρύθμιση, καλύτερη ρύθμιση θέλουμε όλοι. Ακούγοντας τον εισηγητή, ε, πιστεύω ότι έχει τη σωστή προσέγγιση και θα είναι κυλισμένη η έκθεση. Πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Ακόμη και εγώ τα καταφέρω να είμαι ρεαλιστής ενίοτε θα ήθελα να υποβάλω ερωτήματα στους εκπροσώπους της ΑΙΟΣΚΟ και της ΣΥΖΕΡ. Όταν πηγαίνω στην κεντρική τράπεζα της χώρας μου, που και οι αρχαιότερες στην Ευρώπη, μου λένε ότι πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας στη ρύθμιση, στην νομοθετική ρύθμιση για το τραπεζικό τομέα. γιατί λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα στις κεντρικές ε, τράπεζες, ασχολούμαστε με τα πλέον σημαντικά ζητήματα. Εσείς ε, πώς τοποθετήσετε. Ναι μεν ε, ζητούμε ρύθμιση, αλλά χρειάζεται προσωπικό, κατάλληλα καταρτισμένο, με τα κατάλληλα προσόντα για να γίνει αυτό. Και δεύτερον, αυτό το μορατόριο σε τρία χρόνια για τις τρίτες χώρες, αν κατάλαβα καλά, αυτό σημαίνει ότι θα αποκλείσουμε τον υπόλοιπο κόσμο ούτω ώστε να έχουμε περισσότερο κεφάλαιο στην Ευρώπη. Κατάλαβα καλά, μπορείτε να το σχολιάσετε. Όλοι και ο κύριο Γκέμπλε θα συμφωνήσουν ότι χρειαζόμαστε κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόληση. Ε, παρακαλώ σχολιάστε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτάκι. Τα πηγαδάκια έξω παρακαλώ. Κύριε Κάμφερ, Καμφά, ε, ε, δεν θέλετε το λόγο τελικά. Ο κύριος Κλουτ, ένα λεπτό να σε εντοπίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ουσιαστικά έχουμε ακούσει εκπροσώπους των ταμείων. Μόνο δύο συνδικαλιστές που έβαλαν άλλη ε, σκοπιά στη συζήτηση. Στην εκλογική μου περιφέρεια, που είναι η περιοχή Ρούρ και είναι από τα μεγαλύτερα οικονομικά ε, περιβάλλοντα στην Ευρώπη, τα ε, συνταξιωτικά ταμεία επιμένουν στον εξορθολογισμό ε, των υποθυθέμενων των επιχειρήσεων. Οπότε δεν δημιουργούνται θέσει απασχόληση, μάλλον απολύονται εργαζόμενοι, παρόλα όσα λέγουν οι ενδιαφερόμενοι. Εσεί λοιπόν που εκπροσωπείτε τα ταμεία, πώ θα φαντάζεστε όλα αυτά και ποια είναι η θέση σα. Α πούμε στη δική μα περιοχή του Ρουρ, πώς θα απορροφηθούν αυτές οι θέσεις απασχόλησης που χάθηκαν τα τελευταία 10-15 χρόνια λόγω αύξησης της πίεσης για παραγωγικότητα. Θα με ενδιαφέρει η άποψη των ε, οικονομολόγων. Γιατί υπάρχει αυτή η ιστορία των ταμείων που είναι προβληματική για τους εργαζομένους. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ μια πολύ μικρή ερώτηση. Δική μου. Διότι ένας ή δύο μιλητές ε, ανέφεραν την ανάγκη παγκόσμια αντιμετώπισης και πριν από λίγες εβδομάδες μόλις ε, εγώ και άλλα μέλη είχαμε πάει στι ΗΠΑ για να συζητήσουμε τα δικά του ε, θέματα ρύθμιση. Έχουν το ίδιο σύστημα καταχώρηση, αλλά τα μεγάλα συνταξιωτικά ταμεία ε, περνάνε μέσα από το, σύμφωνο, από το Συμβούλιο Σταθερότητα. Συγγνώμη και ε, φαίνεται πολύ ε, αδυσόπιτη ρύθμιση και πολύ ισχυρή και τα περισσότερα συνταξιωτικά ταμεία ε, κανονικά συλλαμβάνονται εντό εισαγωγικών από τα παράγωγα και την ομοθεσία για τα παράγωγα γιατί είναι μεγάλοι χρήστες swap και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα περιορισμού και στην εποπτεία και στη διαχείριση και δεν ξέρω ίσως τα μέλη του πάνελ θα μπορούσαν να σχολιάσουν τις ιδέες του G20 να τις ε, συνδυάσουμε μαζί με την οδηγία και τον κανονισμό για το AIFM και να δούμε όσα γίνονται και στις ΗΠΑ. Θα επανέλθω τώρα λοιπόν στο πάνελ για να μας απαντήσουν το πιο απλό ε, είναι να σας δώσουμε το λόγο με την ίδια σειρά που μιλήσατε προηγουμένως, αλλά παρακαλώ να περιοριστείτε στις απαντήσεις σας σε ερωτήσεις που σας έγιναν άμεσα, διότι έχω περίπου 10 βουλευτές που θέλουν να σας κάνουν ερωτήσεις ε, επιπλέον. Και ο χρόνος τρέχει. Παρακαλώ ένα λεπτό, το πολύ πολύ δύο λεπτά, αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, η Βερένα πρώτη. Sorry. Excuse me. Thank you. Θα ευχαριστώ πολύ και θα προσπαθήσω να είμαι και σύντομη και συγκεκριμένη. Το πρώτο ερώτημα που μου απευθύνθηκε ήταν αν θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στις τράπεζες και στο, στη ρύθμιση των τραπεζών ε, γιατί δεν έχουμε ε, παραπεριορισμένους πόρους αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι σωστό το ότι πρέπει να εστιαστούμε στο τραπεζικό σύστημα και γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτή την οδηγία και έχουμε συνέστηση του προβλήματος. Το θέμα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να προβλέψουμε τους συστημικούς κινδυνούς οι οποίοι μπορεί να προκύψουν μέσα από την, στην αγορά και γι' αυτό ειδικά το θέμα της παροχής πληροφόρησης από τα μία αντιστάθμισης κινδύνου από τους διευθυντές τους θα ήταν ε, πολύ αξιόλογο αυτό, οποιαδήποτε επιπρόσθετη πηγή πληροφόρησης και πιστεύουμε ότι συμφωνώ με αυτό η Κεντρική Τράπεζα για να μπορούμε να απομακρύνουμε τους συστημικούς κινδύνους που προκύπτουν σε άλλους τομείς της αγοράς. Δεν είναι δηλαδή αυτός ένας τομέας στον οποίο πρέπει να επισέλθω. Για τα θέματα των αναγκών των χωρών είναι πολύ σημαντικό από την άποψή μου να υπάρχει κεφαλαϊκή ροή η οποία να δουλεύει ε, για να ικανοποιεί τους ε, καταναλωτές και τους επενδυτές στον κόσμο ολόκληρο και αυτό το λέμε στην εισήγησή μας ε, για τις Ηνωμένε Πολιτείε από ό,τι καταλαβαίνω καταρτίζουν τώρα μια νομοθεσία η οποία θα θεσπίζει τα ταμεία της αντιστάθμισης κινδύνου και θα λέει τι πρέπει να κάνουν οι διευθυντές τους. Ε, εμείς στην ΕΟΣΚΟ θέλουμε να διασφαλίσουμε το ότι θα συνεργαστούμε με τις αρχές της ρύθμισης για να έχουμε μια λογική αντιμετώπιση αυτού του καθεστώτος και βεβαίως συνεργαζόμαστε και με τις ΗΠΑ πάνω σε αυτό ακριβώς το σημείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα, θα ήθελα να πω κάτι για την παρέμβαση του κυρίου Γκέμπελς. Η απάντηση δεν είναι να, μην, να τα αφήσουμε όλα όσοι έχουν και να μην τα ακουμπάμε. Όχι. Χρειαζόμαστε μία αντίδραση στις συγκεκριμένε ανάγκες. Αν έχουμε μεγάλα ε, ταμεία αντισταθμιση κινδύνου πρέπει να εξετάσετε και τους μεγάλους συστημικούς κινδύνους. Ε, το αντίστροφο ισχύει όταν εξετάσετε την περίπτωση των μικρών ταμείων. Για να απαντήσω σε μια άλλη ερώτηση, το ίδιο ισχύει και για τους επενδυτές. Σε κάποια κράτη-μέλη αυτά ισχύουν για τα hedge funds, για τα ασφαλιστικά προϊόντα που διανέμονται στο ευρύ κοινό, χρειάζονται μέτρα προστασίας των επενδυτών. Αυτό δεν ισχύει αν μιλάμε μόνο για μεγάλους θεσμικούς επενδυτές ε, παρόλα αυτά. Δεν είμαι πεπισμένο ότι οι θεσμικοί επενδυτέ είναι σε θέση πάλι να αυτοπροστατευτούν. Ε, και αυτό το δείχνει η εμπειρία μα από το παρελθόν. Κάποιες από μεγάλες επιχειρήσεις, παραδείγματο χάρη, δεν μπορούσαν να αυτοπροστατευτούν με ικανοποιητικό τρόπο. Οπότε χρειάζεται διαφοροποίηση των τεχνικών που χρησιμοποιούμε. Για την κατάχρηση τη θέση στην αγορά είδαμε στη ΣΥΠΑ και γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά ότι αυτό συνέβη. Μια ε, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση κατάχρηση τη θέση στην αγορά. Υπήρξε υπήρξαν υποψίες στο παρελθόν για κάτι αντίστοιχο στην Ευρώπη, αλλά τελικά δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε τους ε, υπόπτους. Ε, ανέκαθεν ε, και ητούσαμε τι εξελίξει στην αγορά, τον όγκο, τι τιμέ κτλ. Αλλά με τι υποψίε που είχαμε δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε του υπόπτου. Τώρα για πρώτη φορά στη ΣΥΠΑ ε, εντοπίστηκαν οι παίκτε, αυτοί που δίνουν τι εντολέ ε, στην αγορά και τελικά ε, πρόκειτο για μεγάλη κατάχρηση και δεν αφορά αυτό μόνο τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου. Δυστυχώς είναι εξαπλωμένο το φαινόμενο και είναι πολύ καλά κρυμμένα αυτά τα ταμεία γιατί λειτουργούν σε έναν αδιαφανή κόσμο οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό που για πρώτη φορά οι ΙΠΑ μπόρεσαν να τραβήξουν αυτό το παραπέτασμα της αδιαφάνειας και να αποκαλύψουν τα όσα συνέβαιναν στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς θα ήθελα να αναγγείλω το θέμα των πιστοτικών οργανισμών του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομίζω ότι δεν θα ήταν πάρα πολλοί που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το θέμα της ευθύνης των θεματοφυλάκων και θα υπήρχε ένα πρόβλημα γενικά με τους ε, επενδυτές. Νομίζω ότι προσωπικά η άποψή μου είναι ότι οι επιπτώσεις για τις αναδιόμενες αγορές είναι κάτι που το σχολίασε και ο συνάδελφος ε, εξάλλου. Η, μέσα στην Ευρώπη και έξω από την Ευρώπη ε, παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον εκεί. Θα υπήρχε μείωση της παροχής ε, υπηρεσιών γενικά και θα είχε αυτό σχέση βεβαίως με τον κίνδυνο, με, το, με την μείωση της ε, ε διασφάλισης από τον κίνδυνο. Ε, και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια εφαρμογή της διασφάλισης του κινδύνου πιστεύουμε και μάλιστα με μεγάλη αυστηρότητα και γι' αυτό ε, εάν το δούμε έτσι είναι πάρα πολύ απλό να καταλάβει κανείς ότι θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος ειδικά σε τομείς όπου είναι υψηλός ο κίνδυνος ε, και πολύ συχνά θα πρέπει να υπάρχει υψηλή επιστροφή του κεφαλαίου απόδοση δηλαδή, δηλαδή όταν υπάρχει ψηλό κίνδυνος. Υπάρχουν όμως ε, ορισμένοι τομεί όπου έχουμε πολύ χαμηλά επιτόκια ε, και εκεί πρέπει να διαχειριστεί κανεί ε, οπωσδήποτε το θέμα του κινδύνου. Ε, το δεύτερο που με ρωτήσατε ήταν σχετικά με τις, ε, τη συνεργασία μεταξύ ΙΠΑ και ΕΕ. Νομίζω ότι βασίζεται ε, σε διάφορες επαφές που έχουμε σε ρυθμιστικό επίπεδο για με το FSA παραδείγματος χάρη που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερος διάλογος και να δαπράττει περισσότερος χρόνος πάνω σε αυτά τα θέματα των συστημικών κινδύνων τα οποία δεν αρνούμεθα ότι υπάρχουν και τα αντιμετωπίζουμε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο ρυθμιστικός διάλογος θα έδινε μια πιο συντονισμένη προσέγγιση αυτών των θεμάτων και βεβαίως και μια καλύτερη ρύθμιση ε, όλων αυτών των ε, ομίλων. Και βεβαίως ε, έχω συνέστηση του θέματος. Ευχαριστώ. Ε, εγώ θα απαντήσω το, ε, στο ερώτημα που τέθηκε σχετικά με τον ε, περιορισμό των παροχιών σε σχέση με την ευθύνη των θεματοφυλάκων. Ε, δείξαν τα στοιχεία που είχαμε πάρα πολύ σαφώς ότι η σωστή διαχείριση του κινδύνου βασίζεται σε μία καλύτερη ε, μεσητεία και θα πρέπει να καταλάβουμε τα προβλήματα τα οποία τίθενται από τα συμβόλαια γιατί νομίζω ότι μία μεγάλη μείωση στους παροχή συγκεντρώνεται σε έναν αριθμό κινδύνων που δημιουργεί ε, ε, έναν μεγαλύτερο κίνδυνο κάτι που είναι αρνητικό για τους επενδυτές. Ευχαριστώ. Το μικρόφωνο. είμαστε κατά ορισμένων πραγμάτων αλλά δεν είμαστε κατά της υποστήριξης της ε, ε, νέας ρύθμισης. Αυτή η ρύθμιση που αφορά τα ταμεία ανταστήθμισης κινδύνων μας βρίσκει πολύ πίσω, 100% πίσω, 100% πίσω στο θέμα της διαφάνειας γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους παραδοσιακούς managers οι οποίοι πρέπει να κατανοήσουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε μια κρίση ε, γιατί στην κρίση κανείς δεν ήξερε πόσο βαθύ ήταν το πρόβλημα στην πραγματικότητα και υπήρχε μια υπερβολή της όλης κατάστασης αλλά τα στοιχεία κλειδιά σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι γίνεται μια σαφής διάκριση γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα του περί τίνος μιλάμε. Γίνεται μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα και υπάρχει ένα overspill σε άλλους τομείς που για μένα είναι σαφές ότι υπάρχει ε, γιατί όλα αυτά τα θέματα ε, πρέπει να πούμε ότι αφορούν αυτό που ονομάζουμε μία εναλλακτική, ένα εναλλακτικό ταμείο επενδύσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ε, κρατήσουμε στο μυαλό μας και μια τελευταία παρατήρηση γιατί και εγώ είχα φτάσει ε, στο όριο και ξέρω πως έχει η κατάσταση που δεν μπορώ να σχολιάσω εδώ αλλά πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή η βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χρηματοδότηση της πραγματικής αγοράς και αυτό ισχύει και θυμάμαι ότι για τις αγορές ισοτιμίες, για τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες δεν επενδύουν στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και αυτό ισχύει τον τελευταίο καιρό τελικά τι θα γίνει, πώς θα περάσουν τα χρήματα μέσα στις ευρωπαϊκές εταιρείες, με ποιο τρόπο. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας σαν ερώτημα. Ευχαριστώ, Κρίστα. Ευχαριστώ. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με τον συνάδελφό μου. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε καθόλου κατά της ρύθμισης. Είμαστε, μιλώντας για τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία, χρειαζόμαστε ρύθμιση. Αλλά το θέμα είναι τι είδους ρύθμιση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις δραστηριότητες των εναλλακτικών επενδυτικών ταμείων. Όχι μόνο την οργάνωση και την οργανωτική δομή, Πρέπει να δούμε τις αμοιβέ, τη μόχλευση, τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται τα επενδυτικά ταμεία. Ο εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου με ρώτησε αν είναι δυνατόν να έχουμε τη ρύθμιση τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν όχι σε παγκόσμιο. Δεν είναι αυτή η βέλτιστη λύση, αλλά από το να το αφήσουμε στην αρμοδιότητα των εθνικών αρμοδίων αρχών ναι, είναι καλύτερο, γιατί θα υπάρξει Ανταγωνισμό, ανάμεσα στα κράτη-μέλη που θα έχουν τα, τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυτά που θα έχουν υψηλότερη ρύθμιση. Αυτό θα επισύρει μεγαλύτερο κόστο και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να είναι ο βασικό αρχιτέκτονας του νέου κανονισμού για τη μόχλευση. Πρέπει να είναι κοινή προσπάθεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κύριε Γκέμπελ, εφόσον μα ζητάτε λύσει και δίκιο έχετε, υποστηρίζουμε ε, την νομοθεσία, αλλά παραδείγματο χάρη για επιμελητή είναι αυστηρότερα τα πράγματα για τα συνταξιδοτικά ταμεία ε, σε, σχέση με τα ε, ενεργά hedge funds. Εμεί δεν επενδύουμε σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και για να ρίχνουμε το βάρο στην μόχλευση και στο φορολογικό αρμπιτράζ. Και με αυτή την οδηγία δεν θα αλλάξει η κατάσταση για τους υπολείπους. Ε, ε, οι λύσεις υπάρχουν ε, στην βιομηχανία, στον κλάδο, σε ορισμένο βαθμό, αλλά όχι όλες. Για τις ομάδες στοιχείων ενεργητικού υπάρχει εξαίρεση για τα συνταξιδοτικά ταμεία μέσα στην οδηγία. Εμείς προτείνουμε να προβλεφθεί εξαίρεση για τα μικρά συνταξιδοτικά ταμεία και τις ομάδες στοιχείων ενεργητικού, pools of assets και υπάρχουν δυσεπίλητα προβλήματα. Χρειάζεται, να, λέγοντας, ε, ε, κλείνω λέγοντας ότι χρειάζεται ρύθμιση για τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία, αλλά το Κοινοβούλιο πρέπει να βρει λύση και να βρει κριτήρια, ούτω ώστε οι ιδιώτες επενδυτές να μπορούν να επενδύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με ασφάλεια. Ευχαριστώ. Yeah, ναι, ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Γκέμπελς. Γιατί χάνονται χρήματα και δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και όπως ε, εξήγησαν οι προαλήσεις, ε, πιστεύουμε ότι χρειάζεται ρύθμιση, όντως, αλλά να ανταποκρίνεται και να απαντά στα πραγματικά προβλήματα. Και αυτό είναι θέμα της μακροοικονομικής σταθερότητας. Εκεί θα πρέπει να εστιαστούμε. Για τα δικά μας συνταξιωτικά ταμεία δεν έχουμε υπερβολική μόχλευση. Δύο-τρεις φορές ε, ε, είναι το μέγιστο. Εμείς είμαστε σε διαφορετική κατηγορία. Ο άμεσος αντίκτυπος της κρίσης αυτής δεν μας έπληξε μας. Δεν είχαμε έκθεση εμείς αυτούς που είχαν πάρει ε, πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Έμεσα όμως έχουμε πληγεί πολύ σκληρά. Και αυτό είναι σημαντικό. Αν δούμε τα τελευταία πέντε χρόνια τι έχουν κάνει τα hedge funds και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι μείον 3 με 5% των επενδύσεων. Οπότε και σε σχέση με την κρίση είναι σχετικά καλή ε, επίδοση. Ε, αν δούμε όμως ε, ε, τι γίνεται με τα ε, κεφάλαια που έχουν χάσει 30 και 40% ε, του χαρτοφυλακίου υπάρχει πρόβλημα και ανησυχία. Και πολλά από τα Ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν πέσει κάτω το 100%, δηλαδή έχουν περισσότερα στοιχεία παθητικού παρά ενεργητικού. Έχουμε λοιπόν καθημερινή αξιολόγηση, καθημερινή εκτίμηση για να δούμε ε, τι γίνεται με την οικονομική ανάκαμψη και ποιες είναι οι συνέπειες για τα κέρδη μας ήδη έχουμε ξεπεράσει το 100%. Δηλαδή έχουμε περισσότερα στοιχεία ενεργητικού παρά παθητικού. Ε, είμαστε στο συν. γιατί ήταν πολύ χαμηλά τα επιτόκια. Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και η Αμερικανική ε, Federal Reserve είχαν πολύ χαμηλά επιτόκια και πολύ απαραίτητα για να ξεπεριστεί η κρίση. Χρειάζεται βεβαίω ε, ρύθμιση και νομοθεσία, αλλά να επικεντρώνεται στου πραγματικού κινδύνου που είναι στον τραπεζικό κλάδο, όπω είπε ο κύριο ε, Σμιτ. Είχαν τεράστιου κινδύνου, έκαναν τεράστια μόχλευση και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει του πολιτικού και να ρυθμιστούν όλοι, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα συνδικάτα έχουν ορισμένα σχόλια να θέσουν. Παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο σύντομα για το σχόλιο που έθεσε ο κύριος Κρύφη για αυτούς τους τομείς ένα γενικό θέμα καταρχήν ότι σε όλες ε, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες υπάρχει το, τίθεται το θέμα των συστημικών κινδύνων που δεν καλύπτονται. Ε, πιστεύουμε ότι αυτά απευθύνονται και στην πραγματική οικονομία και ότι υπάρχουν ορισμένοι τομείς κλειδιά και ιδίως όταν συζητάμε ε, το θέμα της μόχλευσης και ποια πρέπει να είναι. Ε, είναι βασικό ότι δεν είναι απλώς το θέμα η χρήματο-οικονομική σταθερότητα και η συστημική κίνδυνη αλλά και το πρόβλημα της πραγματικής οικονομίας η οποία έχει μια πολύ υψηλή μόχλευση ε, και εδώ ε, επισέρχεται και το θέμα των εργαζομένων σε αυτές τις εταιρείε. Έκανα ένα σχόλιο προηγουμένως για τις ανάγκες της ποικιλομορφίας που πρέπει να υπάρχει για να υπάρχει καλύτερη απόδοση στα επιτόκια ε, για την ανάκαμψη της οικονομίας η οποία πρέπει να προέρθει για όλους μας χρειάζεται ε, αυτή η ανάκαψη του χρηματοοικονομικού τομέα και αν υπάρχει οποιαδήποτε επιτυχία σε αυτό το τομέα κλειδιά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της οικονομίας και αυτό είναι το θέμα που θέτει και αυτή η οδηγία σε σχέση με την μόχλευση αλλά πρέπει οπωσδήποτε και να προστατεύονται καλύτερα τα συμφέροντα των εργαζομένων. Ε, ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στους επόμενους ομιλητές. Λόγω του χρόνου ε, θα έπαιρνα όλους τους υπόλοιπους βουλευτές τις ερωτήσεις που ενδεχομένως θα ήθελα να θέσουν. Έχω λοιπόν έναν κατάλογο των εξής. με αυτήν τη σειρά που του διάβασα τα ονόματα η Προεδρεύουσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απάντησαν ήδη οι πυρογνώμονες. και είπαν ότι θέλουμε να ε, έχουμε περισσότερη διαφάνεια, ανατολισμό στο συστημικό κίνδυνο, μεγαλύτερη ενημέρωση. Ο κ. Μπούρμαν μίλησε και για τη συμπεριφορά και κανόνες που πρέπει να διέπουν. Εμείς είμαστε νομοθετικό σώμα εδώ μαζί με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο ακόμα δεν έχει πει τίποτα. Έχει πει όμως κάτι η Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία έχει καταθέσει πρόταση στα εξή τέσσερα σημεία. Σαφώς στενότερα πεδία εφαρμογής, όχι πλέον διαχειριστές, managers του, του, των ταμείων, αλλά πιο περιορισμένοι με ε, ανάθεση, με τραπεζικές εγγυήσεις μέχρι 50%, χωρίς ανώτατο όριο στη μόχλευση και λιγότερη ενημέρωση για την επιρροή και για ε, το μοχλό. Και γιατί αυτή η πρόταση ενδείκνυται καλύτερα για την αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου από ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τη δική μου πολιτική ομάδα, αυτό δεν συνιστά πρόεδρο. Μπορείτε να μας ε, εξηγήσετε γιατί αντιμετωπίζετε καλύτερο συστημικός κίνδυνος με αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές και ε, τη μονάδα πολιτικής που μας ε, έδωσε τα στοιχεία για να προετοιμαστούμε. Εγώ θέλω να αναφερθώ στα θέματα μόχλευσης και στις τρίτες χώρες. Ε, αν μπορούσατε να μου απαντήσετε για τη μόχλευση στα επενδυτικά κεφάλαια υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές για τη μόχλευση και μπορούμε να έχουμε νέα μέτρα. Νομίζω ότι αυτό να μην είναι το καλύτερο. 70% των στοιχείων ενεργητικού στα ευρωπαϊκά εναλλακτικά ταμεία ε, υπάρχει μόχλευση μία και δύο φορές περίπου. Ε, πώς ελέγχεται αυτό και πώς είναι προσβάσιμο σε ε, όλα τα παιδιτικά κεφάλαια ε, και ε, στη μεσητεία, στο brokerage. Και το δεύτερο Ακούσαμε ότι το 94% των στοιχείων ενεργητικών, των συνταξιωτικών ταμείων έχουν την έδρα τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε ο ότι είναι σημαντικό ε, να διαβάσουμε ένα κείμενο FSA του Οκτωβρίου που λέει ότι 35% ε, των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 90% του κεφαλαίου κινδύνου τελικά μπορεί να διαφεύγει ε, ε, των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Πώς μπορείτε αυτό να το σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Θέλω να σας θυμίσω να μην μιλάτε τόσο γρήγορα. Ανάβουν κόκκινα φωτάκια εδώ, λαμπάκια. Δεν σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Υπερβάσου. Ευχαριστώ. Η καλύτερη νομοθεσία μας είπανε θα γίνεται μέσα στο σκοτεινό θάλαμο. Εγώ άλλη συζήτηση εκτός από τη δημοκρατική δεν γνωρίζω. Και όταν μιλάμε για τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία, τα κερδοφόρα ταμεία μου λένε είναι απαραίτητα για την οικονομία. Ναι, αλλά όταν έχουν αναπτυχθεί εκθετικά και όταν δεν υπάρχουν επενδύσεις είτε από κρατικής πλευράς είτε από ιδιωτικής πλευράς δεν νομίζω ότι ισχύει. Δύο ερωτήσεις. Ε, ακούσαμε ότι δεν χρειάζεται να επιβάλλουμε υποχρεώσεις ε, στις διαχειριστές ε, των hedge funds σε σχέση με αυτές που ισχύουν για του διαχειριστές των ΟΣΕΚΑ. Ε, ναι, αλλά ούτω ή άλλω χρειάζεται ρύθμιση και στου ΟΣΕΚΑ. Α αρχίσουμε με τα hedge funds που μα απασχολούν τώρα και μετά. Ε, παρόδο θα διορθώσουμε την κατάσταση και στους ΟΣΕΚΑ. Γιατί Ξέρετε ότι υπάρχει το πρόβλημα των θεματοφυλάκων και για τους ΟΣΕΚΑ και ας μην προ... Ε, προβάλλουμε αυτό το επιχείρημα ότι πρέπει να αρχίσουμε πρώτα από τους ΟΣΕΚΑ. Το θέμα του θεματοφύλακα πρέπει να μα απασχολήσει και στις ε, δύο περιπτώσεις. Για την διακυβέρνηση μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Ποια είναι τα τρία-τέσσερα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για τη διακυβέρνηση, η αμοιβή των στελεχών. Ναι, είμαι σίγουρη ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να ρυθμίσουμε. Αλλά υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Και τώρα, ε, δεν θέλω να μιλάμε για τη ρύθμιση των hedge funds, για τη ρύθμιση των προϊόντων, ε, η απαγόρευση των ακάλυπτων πωλήσεων, το short selling. Τι έχετε να πείτε για αυτό το θέμα. Χρειάζεται η απαγόρευση για τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία, ε, η απαγόρευση των ακάλυπτων πωλήσεων. και ο εκπρόσωπος της ΣΥΖΑΡ που μας είπε ότι δεν τον αφορά το θέμα θα ήθελα να μου πει Συγκεκριμένα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θεωρείτε ότι ανάμεσα στο hedge funds και στους εποπτικούς μηχανισμούς που θεσπίζουμε τώρα πρέπει να υπάρχει μια γέφυρα. Τι πρέπει να περιμένουμε την επόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για να φτιάξουμε αυτή τη γέφυρα. Αυτό πρέπει κανονικά να μπορεί να γίνει τώρα όπου και αν έχουν φτάσει οι εργασίες στο Συμβούλιο. ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω σύντομες ερωτήσει στους εμπειρογνώμονες μας. Πρώτον, κυρία Βός, νομίζω ότι όλο αυτό το θέμα για τις τρίτες χώρες, την αντιστοιχία κτλ. Είναι δύσκολο να ε, ρυθμιστεί, να υπάρχει παγκόσμιο συντονισμός και παγκόσμιες προδιαγραφές. Εγώ ανησυχώ, όπως και άλλοι, ότι εσείς μιλάτε πολύ για προσέγγιση αρχών και έτσι λειτουργείτε, αλλά υπάρχουν κάποιοι τομείς στην τράπεζα, ας πούμε, και στην οδηγία αυτή που ε, προσέγγιση είναι περισσότερο βάσει των κανόνων, όχι παγκόσμια, όχι συνολική. Πώς συνάδουν αυτά, πώς συνδυάζονται τα δύο. Αν δεν υπάρχει παγκόσμια συμφωνία θα έχουμε επιπτώσει για τις τρίτες χώρες. Και όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στα hedge funds, στις εγκρίσεις ας πούμε, στις ε, ε, καταχωρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Οπότε θέλω να μάθω ποιες είναι οι ιδέες σας και οι απόψεις σας για αυτό το θέμα και ένα σύστημα αρχών ε, πώς εφαρμόζεται αν δεν βασίζεται στους κανόνες. Καλές οι αρχές, αλλά πώς θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν, να συμμορφωθούν. Στη συνέχεια, όταν κάνετε επενδύσεις, Πώ θέλετε να ρυθμίζετε από την νομοθεσία. Και τον κύριο Ντούμα θέλω να ρωτήσω. Είπατε ότι έχετε αυστηρού κανόνε για τι επενδύσει σα Και πάλι να σα ρωτήσω, ποια είναι τα στοιχεία ε, δημοσιότητα στην οδηγία θα σας βοηθήσουν για να έχετε καλύτερη κρίση και καλύτερη απόφαση. Γιατί βλέπουμε πώς αυξάνονται οι επενδύσεις ε, στα hedge funds. Στο Ηνωμένο Βασίλειο από 5% έχει φτάσει στο 30% και ακούμε και μέχρι και 75% των συνταξιδοτικών ταμείων θα επενδύουν σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου. Και ε, τέλος, είπατε ότι δεν είστε από τη σχολή που δεν θέλει κανόνες ε, και ε, θέλουμε και εμείς να διδαχθούμε από τη δική σας πραγματογνωμοσύνη. Αλλά αν θέλετε ε, να ονομάζεται τις περιπτώσεις αυτές μπλήψη, δεν ξέρω πόσο, από το 1998 μια εταιρεία κατέρευσε όταν δανείστηκε 120 δισεκατομμύρια δολάρια ε, σε μια επένδυση 4,5 εκατομμύρια σε δύο μέρες έχασε το 90% Πού ήταν τα στοιχεία ενεργητικού, από πού προήλθαν από επενδυτικέ τράπεζε και συνταξιωτικά ταμεία και εξατμίστηκαν. Τι γίνεται λοιπόν, πού είναι ο συστημικό κίνδυνο, ακόμα και αν ένα μπλίπι, όπω λέτε, ή κάτι άπαξ και μετά δεν επαναλαμβάνεται. Άμα χαθούν τα λεφτά, τι γίνεται. Um, Ευχαριστώ. Θέλω να ασχοληθώ με τις συντάξεις. Όπως ε, έχουμε συζητήσει και σε άλλες επιτροπές, ε, το αυξανόμενο χάσμα στις συντάξεις και το ότι Καλό είναι που ζούμε όλοι περισσότερα χρόνια, αλλά έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και αυτό συνειδητά πρόκληση για όλους. Και άρα όλοι ή θα πρέπει να εργαζόμαστε όλοι για περισσότερο χρόνο ή να παίρνουμε λιγότερα λεφτά στη σύνταξή μας θα είναι πολύ δυσκολότερο για τα συνταξιδοτικά ταμεία στην Ευρώπη να επενδύσουν εκτός Ευρώπης ή εναλλακτικά θα ε, είναι πολύ πιο δύσκολο να έχουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού ανάμεσα στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ταμεία εκτός Ένωσης. Παραδείγματος κάνει αν ισχύει λόγος για τη μόχλευση εδώ και όχι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους διαχειριστές τώρα, αν κατάλαβα καλά, όταν μιλάμε για τους μεγαλύτερους διαχειριστές δεξιδοτικών ταμείων, δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν επενδύσεις στα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία και αν ναι, αν ήμασταν ένας από τους συνταξιούχους σας Πόσα θα έχουμε χάσει φέτος από τη σύνταξή μας ε, λόγω αυτών των επενδύσεων. Τι κοστίζει στο ταμείο σας ε, σε κάθε συνταξιούχο το ότι δεν μπορείτε να επενδύσετε σε, αυτούς, ε, σε αυτά τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία. Πρόεδρος, η Ελίζα Φερήρα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να θίξω αυτά τα θέματα που έθιξε η συναδελφός μου. Εμένα με απασχολούν δύο θέματα. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία τα οποία θεωρούνται ως ε, ζωτικού συμφέροντος για να μπορέσουμε να δώσουμε το ίδιο νόημα σε αυτό που λένε οι πάντες ότι χρειάζεται μια καλύτερη οδηγία. Τη χρειαζόμαστε αυτή την οδηγία. Οπότε τι συστάσεις κάνετε πάνω στα πολύ σοβαρά θέματα που είναι η μόχλευση, ευθύνη των ε, θεματοφυλάκων, ο συστημικός κίνδυνος Πρέπει να δούμε τα γενικά προβλήματα τα οποία καθορίζουν τα πράγματα. Πρώτον. Δεύτερον, ε, μου έκανε, ανησύχησα πάρα πολύ, μου έκανε εντύπωση ότι ε, όταν άκουσα τον κύριο Βάιμα, ο οποίος ε, είπε ότι μιλούσε για την προσωπική του γνώμη. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα είναι σημαντικό και θεωρώ ότι όλα τα θεσμικά όργανα που δουλεύουν ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό το θέμα καθώς και το διεθνές πλαίσιο πρέπει να εστιαστούν πάνω σε κοινού κανόνες. Πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο κοινό το οποίο δεν το έχουμε για να μπορέσουμε να ασκήσουμε μια κριτική πάνω σε αυτή την πρωτοβουλία γιατί εδώ μιλάμε για τη δημιουργία ενός ανισότιμου πεδίου ε, στην Ευρώπη. Μπορείτε λοιπόν να μας προσδιορίσετε ε, τι είναι ο, πιο είναι ο της Ευρώπης και ποιο είναι ο ρόλο αυτών των διεθνών οργανισμών οι οποίοι να αναλάβει τη δέσμευση να δημιουργήσουν ε, νέους κανόνες αγοράς. Ε, ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να εργαστούμε. Ευχαριστώ. Εγώ έχω δύο πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Το πρώτο ε, αφορά τα ταμεία τα συνταξιοδοτικά και αυτούς που τα εκπροσωπούν. Καταρχήν τι απώλειες είχαν οι εργαζόμενοι της Ευρώπης οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι κατά τη διάρκεια της κρίσης σε συνταξιοδοτικά ταμεία, πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα προς τα συνδικάτα. Το Ευρωπαϊκό Σύμβουλο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας καλούν να σκεφτούμε πάνω τη, στη στρατηγική της Λισαβόνας 2 για μια μεταρρύθμιση των ε, συντάξεων. Εσείς μιλάτε για κεφαλαιοποίηση, πρέπει να δώσουμε βάση στην κεφαλοποίηση ή στην ε, ε, κατανομή που είναι μια διαφορετική αρχή η οποία πρέπει να να αναδιανομή, με συγχωρείτε, την οποία πρέπει να αναπτύξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Όπως και πριν θα ακολουθήσουμε την ίδια σειρά μας δώσουν άλλα 5 λεπτά οι διερμηνείς. Αλλά έχετε περίπου ένα λεπτό έκαστος για τις απαντήσεις. Θα υπάρξουν και συμπληρωματικές ενδεχομένω απαντήσεις, αν διατίθεστε. Και υπάρχει και το σεμινάριο, το εργαστήρι, σήμερα το απόγευμα, στο ίδιο κτίριο, στον τέταρτο όροφο, στο 4, στην αίθουσα 4Β1. Λοιπόν, απαντήσεις. Ε, Ρίνα, τελευταίος γύρος απαντήσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε από την δική μας την οπτική γωνία καταφέραμε να συμφωνήσουμε επί γενικών αρχών για τα κοινά σημεία για την νομοθετική ρύθμιση. Φυσικά δεν ισχύουν τα ίδια όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπάρχει συνθήκη, δηλαδή υπάρχουν όρια σχετικά με τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι σημαντικό να έχουμε ελάχιστα πρότυπα ε, με που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις διεθνείς και από τις εθνικές αρμόδιες αρχές όταν διαμορφώνουν τα δικά τους ρυθμιστικά συστήματα για να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται συνοχή ε, αλλά φυσικά οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα αποφασίσουν για τα μεμονωμένα πρότυπα σε επίπεδο κράτους μέλους. Ε, για την εφαρμογή τώρα υπάρχουν ε, ε, εταιρικές ρυθμίσεις για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατάξεων και γίνονται σχετικές εργασίες και στην ΑΙΟΣΚΟ και στη ΣΥΖΕΡ είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τη συνεργασία ούτω ώστε οι κανόνες στους οποίους θα καταλήξουμε να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Χρειάζεται στενή συνεργασία. Έντι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα αρχίσω από τις τελευταίες ερωτήσεις. Όντως, και εμένα με προβληματίζει στη σημερινή συζήτηση. Εγώ ως εκπρόσωπο της, Caesar σας είπα δεν έχω καμία ενημέρωση για το τι συμβαίνει σε επίπεδο συμβουλίου δεν συζητείται. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή δεξαμενή προβληματισμού think tank ε, και θα ήταν ε, χρήσιμο να υπάρξει ένας τέτοιος όμιλο μεταξύ ορισμένων που είναι πολύ καλά πληροφορημένοι και μέλη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ένα όμιλο προβληματισμού, ένα think tank για να προετοιμάσει ένα κείμενο. Τώρα βλέπουμε το ακριβώ αντίθετο. Αύριο, α πούμε, θα έρθουν οι νέε προτάσει, θα δημοσιευθούν οι νέες προτάσεις της Σουηδικής Προεδρίας το μόνο κείμενο που έχω στα χέρια μου είναι αυτό που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στις διαδικασίες. Δεν απόκειται σε μένα να το επικρίνω εγώ. Απλώς σα λέω ότι εδώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου. σα το είπα και προηγουμένως. Γι' αυτό το λόγο και η ΣΥΖΑ δεν ασχολείται και δεν αναφέρεται στι προτάσει εξ όσων γνωρίζω. Ε, μελλοντική αρχή θα πρέπει να υπάρξει μια ανάθεση κάποιων τεχνικών θεμάτων, ας πούμε, Πόση ενημέρωση θα πρέπει να υπάρχει και αποκάλυψη. Τι γίνεται με τη μόχλευση. Ε, αυτά θα πρέπει να τα ε, πούμε σε λεπτομέρειες, όχι σε επίπεδο 1 ή 2, αλλά και σε πιο τεχνικό ακόμα επίπεδο, με προδιαγραφές που θα εκπονήσουμε. Ωραία. Αυτό το είπα τώρα. Άλλο. Ε, για τις ιδέες της Περβάνς Μπερές. Η πρόταση για το θεματοφύλακα ήταν να ισχύει παντού το ίδιο καθεστώς. Όχι όμως το καθεστώς που προτείνεται τώρα, ε, στην οδηγία για τα επενδυτικά κεφάλαια, αλλά για ε, τη ε, δέουσα επιμέλεια, due diligence, για τη διαχείριση, διακυβέρνηση. Δεν συζητήθηκε αυτό σε λεπτομέρειες, αλλά είναι τεράστια ζητήματα αυτά και σε επίπεδο ε, ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και στη σχέση ε, με τις ε, εταιρείε που επενδύονται και υπάρχουν και θέματα ακτιβιστών επενδυτών. Κάποιος το είπε αυτό ο πρόσωπος της Allianz. Τι είναι αυτό το πράγμα, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει activist investors και, και πώς έχουν αναπτύξει αυτή τη δραστηριότητα οι επενδυτές. Το ίδιο ισχύει και με το empty voting. Μου έκανε εντύπωση που αναφέρθηκε και αυτό εδώ, εν πάση περιπτώσει. Ε, για την ε, πώληση ε, αντικρίσματος, το short selling, αυτό είναι ένα δεύτερο στάδιο ε, που πάει και στη διαδικασία επίλυση διαφορών κανονισμών θα πρέπει να γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Δυστυχώς σήμερα παίρνει τρει ημέρε για να γίνει αυτό. Σε κάποιε αγορές γίνεται την ίδια μέρα η ε, επίλυση της διαφοράς ο διακανονισμό. Και στην αγορά αυτή των ε, μετοχών ε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα έπρεπε, αν γινόταν την ίδια μέρα ή σε λιγότερο από τρει μέρες, θα λύναμε και το πρόβλημα του short selling, της πώληση ανεφαντικρίσματος. Ρόμπιν το, θα απαντήσω άμεσα στην ερώτηση της κυρίας Χάπη ποιε είναι οι προδιαγραφές τις οποίες αναζητούμε και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με την οδηγία. Ε, με τα μιλώ, χρησιμοποιούμε διάφορα συστήματα τα οποία βασίζονται ε, στο καθεστώς το οποίο χάσαμε δυστυχώς ε, γιατί υπήρχε μια παράληψη και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα μέσα από το δίκτυο και έχουμε το ε, διάφορους πράκτορες απκάστητη οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ε, είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης και είναι ενδιαφέρον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, τις επόμενες μέρες θα συζητήσουμε με την FSA για να εκπονήσουμε μια κοινή άποψη. Πιστεύουμε ότι η FSA αποφάσισε σωστά να εξετάσει αυτά τα θέματα και να δει τα προβλήματα του, της ροής που προκύπτουν παρόλο που δεν έχει γίνει σωστή θέσπιση μέσα από την οδηγία. Επίσης ε, ε, υπάρχει διαχωρισμός του ενεργετικού ε, και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει μια αναφορά στην, στη ΣΥΠΑ για τα αμοιβαία κεφάλαια και όλες αυτές οι πλευρές είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί και είναι, έχουν κάποια σχέση με την οδηγία και νομίζω ότι θα βοηθήσουν την εξέλιξη μιας καλύτερης διατύπωσης της οδηγίας και θα είμαι πολύ ευτυχής αν μπορώ να συμβάλλω ε, μέσα από αυτό το δίκτυο στην εξέλιξη. Ε, ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση τώρα που έχει ε, σχέση με τους συστημικούς κίνδυνους, τη μόχλευση ε, και τα θέματα τα οποία έχουν σχέση σχέση με την διάσταση εκτός ε, ε, σε σχέση με τους συστημικούς κινδύνους. Ε, καταρχήν σε σχέση με την ε, διαχείριση των Ταμείων Αντιστάθμισης Κινδύνων έχουμε τα μόνο έξι ταμεία τα οποία μπορούν να αποπληρώσουν γιατί υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι οι οποίοι ε, δεν μπορούν να καταμετεθούν. Υπάρχει ε, μία μόχλευση του σε σχέση με τον υψηλό κίνδυνο, κίνδυνο ε, και επίσης η αντιστάθμιση κινδύνου αυξάνει τη μόχλευση και υπάρχει σωστή στόχευση γιατί μόνο με τη σωστή στόχευση του σωστού πράγματος μπορούμε να προχωρήσουμε και να έχουμε μία γενική θέση γιατί αν δεν υπάρχει μία γενική θέση τότε υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος και ε, γίνονται επενδύσεις εκτός ε και εκτός αυτού του πεδίου ε, πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια διαφάνεια ε, για τις, να αντιμετωπιστούν οι συστημικοί κίνδυνοι και ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα είναι ε, η σωστή αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων. Μας ρωτήσατε ποιες είναι, ποια είναι τα θέματα κλειδιά. Ε, εγώ θα ήθελα να σας απαντήσω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες ερωτήσεις και εστίαση στα ε, σωστά προβλήματα. στην Γερμανία είχαμε ένα πρόβλημα με τις ασφάλειες ζωής και είναι κάτι το οποίο αντιστοιχεί με τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι επαρκές το επίπεδο αυτό αν χρειάζεται μια σωστή πρόβλεψη για, την, ε, ε για τους ηλικιωμένους για την ε, τρίτη ηλικίου. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια σωστή πρόβλεψη για τα ε, γεράματα των ανθρώπων που είναι ασφαλισμένοι σε αυτές τις εταιρείες αλλά χρειάζεται ε, μία ε, αντιμετώπιση της, ε, των επενδύσεων και δεν θα πρέπει να έχουμε ένα συνολικό παγκόσμιο επίπεδο στο οποίο υπάρχουν ορισμένοι όμιλοι οι οποίοι διαχειρίζονται τους κινδύνους. Βεβαίως διαχειριζόμαστε τους κινδύνους σε καθολικό επίπεδο αλλά υπάρχουν σε διάφορους τόπους, διάφορες μονάδες που καθιστούν τα πράγματα δυσχερή γιατί πρέπει να εξηγήσουν σε επίπεδο ομίλου τι κάνουν και αυτό είναι ε, τελικά κάτι που φέρει όφελος ε, συνολικά στους επενδυτές ε, σε τελική ανάλυση. Ευχαριστώ. Καταρχήν τα τελευταία χρόνια, που, τα τελευταία ένα με δύο χρόνια όπου υπάρχει επηρεασμό όλων των αγορών που έχουν υποστεί ε, όπως ε, ε, και ε, οι προηγούμενες τα προηγούμενα χρόνια συμβαίνουν τα ίδια πράγματα. πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό και γιατί είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την οδηγία και γιατί είναι σημαντικό να έχουμε καλύτερη διαχείριση του κινδύνου από τα συνταξιοδοτικά ταμεία. δεν νομίζω ότι πρέπει να το συζητάμε αυτό το θέμα. Επίσης η ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους ανθρώπους που έχουν μια σύνταξη είναι μια ποικιλομορφία του πορτφόλιου. Εμείς έχουμε ε, μια καλύτερη διαχείριση των ποσοστών των χρημάτων των κεφαλαίων ε, σε διάφορους τομείς. Επίσης στα κεφάλαια venture, ε, στα startups, στους τέκνοστάτες προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις εταιρείες να αυξηθούν, να αναπτυχθούν και υπάρχουν πολλά τομεία μέσα στην βιομηχανία των εναλλακτικών επενδύσεων που έχουν τεράστια ε, ωφέλη για τις διάφορες εταιρείες και για την κοινωνία γενικότερα. Ζητάμε να έχουμε μια διαφάνεια, θέλουμε μια διαφάνεια πάνω ε, στο θέμα της μόχλευσης και σε άλλα θέματα πολλά, αλλά το κύριο σημείο που μας απασχολεί εδώ είναι ε, γιατί χρειάζεται η διαφάνεια για να μπορέσουμε να έχουμε ε, εκπληρώσει το στόχο της οδηγίας και εμείς σαν επενδυτές μπορούμε να ζητήσουμε πάντα περαιτέρω διαφάνεια γιατί εάν δεν έχουμε επιπρόσθετη διαφάνεια τότε δεν θα κάνουμε επενδύσει. και αυτό είναι ένα πολύ καλό επιχείρημα για αυτούς που θεσπίζουν την οδηγία σε αυτά τα θέματα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι το short selling ε, ε, πρέπει να συνδυάζεται με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρνητικά σχόλια ε, ε, τα οποία απευθύνουν προς το κοινό και μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση μιας ε, εταιρείας. Θα πρέπει αυτό να συνδυάζεται με διάφορες άλλες δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Γιάρτο, ευχαριστώ πολύ. Τρεις ερωτήσεις ήταν προς εμένα. κυρία Μακάρθη με ερώτηση για το ITCM. οι απώλειες δείχνουν ότι χρειάζεται διαφάνεια για τους επόπτες για να μπορούν να ε, εκτιμούν τα θέματα σταθερότητας. Εμείς στις κάτω χώρες έχουμε τα συνταξιωτικά ταμεία που υπάγονται σε αυτούς τους κανόνες. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί κίνδυνος πέρα από κάποιο βαθμό. Υπάρχουν ήδη όρια και μέχρι ένα ορισμένο ποσοστό επιτρέπεται να επενδύουμε σε hedge funds, σε κεφάλαια κινδύνου άλλα. Υπάρχει αυτό, ισχύει. Τώρα, τι αντίκτυπο θα είχε όλο αυτό το εγχείρημα για το κόστος και τους μελλοντικού συνταξιούχους. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί. Και ζητώ ένα πραγματικό έγγραφο, μια μελέτη ενδεικτή που τώρα εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό, προσπαθήσω. Θα πρέπει και ο νομοθέτης ε, να θεωρεί κανονική απόδοση επενδύσεων 6 με 7%. Αυτό είναι ο κανόνας τα τελευταία χρόνια. Αν δούμε το κόστος συμμόρφωσης ποιο είναι και ο κίνδυνο που είναι περιορισμένο. Αυτή η οδηγία δεν περιορίζει το δικό μας κίνδυνο, αλλά για τους μικροεπενδυτές ε, λιανική. Αν θέλουμε να περάσουμε σε 5 με 6%, δηλαδή να μειωθεί η απόδοση κατά 1%, αυτό ε, θα έχει επιπτώσεις 15 ε, με 20% στα κόστος που πρέπει να πληρώσουν οι συνταξιούχοι και τέτοιες περιόδους τώρα μετά την κρίση τι κάνουμε ε, για τους εργαζομένους στην Ολλανδία, γιατί είμαστε κάτω του 100%. Τώρα περιορίζουμε τη διόρθωση του ε, πληθωρισμού. Δηλαδή δεν πέφτουν οι συντάξεις, ε, ε, δηλαδή τις ίδιες συντάξεις παίρνουν ε, στον λογαριασμό του συνταξιούχοι, αλλά δεν τους δίνουμε άτα. Είχαμε 0,7% χαμηλό πληθωρισμό. εντάξει, μέχρι να φτάσουμε στο 130% κάλυψη θα ακολουθούμε να μην δίνουμε αυξήσεις ε, τη μαριθμική ε, αναπροσαρμογή στι